Okay, Jackie, we'll start. Τζάκι, ξεκινήσουμε. Φράγκα, έχει το λόγο. Eurocontrol. Thank you. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλου. Σας ευχαριστώ που δίνετε στο Eurocontrol και σε μένα, με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας ε, σήμερα το απόγευμα την πορεία των πραγμάτων σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, αλλά και τις περαιτέρω εξελίξεις ε, σε ό,τι αφορά το Eurocontrol ε, και στο παρόν και στο μέλλον. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο για να έχουμε και κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο Eurocontrol στηρίζει ενεργά τον, ενιαίο, τον ευρωπαϊκό ενιαίο ενέργειο χώρο και στο παρελθόν εργαστήκαμε σκληρά για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Θεωρούμε ότι το Single European Sky είναι το μέλλον ε, της ε, διαχείρισης της νερές κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και όχι μόνο για τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για όλα τα μέλη του Eurocontrol που σύντομα θα αγγίξουν τα 40 μέλη με την προσχώρηση της Γεωργίας την 1η Ιανουαρίου 2015. Ένα κύριο στοιχείο του Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου, η ουρανού, ε, είναι ο διορισμός ε, της Eurocontrol ως ε, διαχειριστής δικτύου Network Manager. Καταφέραμε έτσι να λειτουργήσουμε πιο γρήγορα για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων και έχουμε μετρήσιμα και αυτά αποτελέσματα. Έχουμε περικόψει και τις δαπάνες μας ουσιαστικά ούτως ώστε να είμαστε τώρα σε θέση να συμβάλλουμε στην περίοδο αναφοράς και τον ε, στόχο επιδόσεων της ε, περίοδου αναφοράς 1. Ε, και αναλογικά μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και για τους στόχους αποδοτικότητας. Επομένως, αν όλα πάνε καλά, όλοι οι φορείς θα κάνουν κάτι αντίστοιχο και αν όλοι καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους, να κάνουν περικοπέ και το καθεξής, θα πετύχουμε τους γενικότερους μα. στόχου μας. Δεν είναι εύκολο βεβαίω, αλλά είναι εφικτό. Βλέπουμε τώρα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα κρατημέλη ε, να ε, μειώσουν τις δαπάνες τους. Για παράδειγμα, μέσω κάποιων υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο ή κάποιες κεντρικές υπηρεσίες σε πιο κεντρικό επίπεδο. Σίγουρα γνωρίζετε τα όσα αναπτύσσουμε με τα κράτη-μέλη και τα ENSP, το στρατό, τα αεροδρόμια, ε, τους ε, διαχειριστές δικτύου των ε, αεροδρομίων και το καθεξής τους τελευταίους μήνες. Ουσιαστικά μιλάμε για 80 ε, υπηρεσίες στήριξης ATM με νέα ουσιαστικές υπηρεσίες, τις οποίες θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά και με χαμηλότερο κόστος, με, με μια πιο κεντρική διάσταση, χωρίς βεβαίω όλα να τα αναλαμβάνει ο Eurocontrol, ούτε να περνάνε ως υπηρεσίες ε, που παρέχονται στον ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, το νέο Caesar σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη βασίζεται γύρω από τις τροχές τεσσάρων διαστάσεων. Επομένω, ένα αεροσκάφος το οποίο έχει ως στόχο να ε, ακολουθήσει μια τροχιά λέει πόσο και θα γίνει αυτό, σε ποιο ύψος και σε κάθε χρονική στιγμή. Αυτές οι πληροφορίες μετά ε, στέλνονται παντού σε όλους ε, τους φορείς και είναι ακριβώς πολύ σημαντική αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτή η ενιαία υπηρεσία για τον σχεδιασμό και την περιγραφή της ε, τροχιά, θα σημαίνει ότι οι πληροφορίες ε, είναι απολύτως συναφείς και συμβατές. Και έτσι αυτό θα μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα σε όλη την Ευρώπη αν σκεφτούμε βεβαίω ότι έχουμε και ε, στρατιωτικά αεροδρόμια. Ανεβαίνει πολύ ο ρυθμός των αεροδρομίων. Πρέπει μετά να σκεφτούμε και το περιβάλλον, γιατί έχουμε και στόχο την μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης καυσίμου. Και πρέπει να δούμε αν ακριβώς θα επιτύχουμε αυτούς τους ε, στόχους ε, για το περιβάλλον. Έχουμε επικεντρωθεί στις υπηρεσίες δεδομένων, γιατί εκεί θεωρούμε ότι η κεντρική διάσταση και προσέγγιση είναι πιο συναφής. Και μάλιστα σε όλες τις συζητήσεις, ε, συνεδριάσεις, εργαστήρια επ' αυτού του ζητήματος που κάναμε τους τελευταίους 12 μήνες, ε, δύσκολα μπορούμε να σκεφτούμε μια φορά όπου κάποιος ξέφρασε αντίθεση με αυτή την ε, κεντρική προσέγγιση των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας στηρίζει ιδιαίτερως και θα επανέλθω στην Κομισιόν και στο SES2 στη συνέχεια. Πού βρισκόμαστε τώρα σε ό,τι αφορά αυτές τις κεντρικές υπηρεσίες. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν αυτή την έννοια συνεργασίας για κάθε μία από αυτές τις κεντρικές υπηρεσίες, οι κεντροποιημένες υπηρεσίες. Ε, ε, οργανώσαμε πάνω από 20 εργαστήρια με όλους τους ενδιαφέρομενους φορείς. Έχουμε απευθυνθεί σαν εξάρτητη εταιρεία για να κάνει την αξιολόγηση ε, κόστους-οφέλους την πραγματοποίησαν και μας είπαν ότι είμαστε αρκετά συντηρητικοί μάλιστα, απεσιόδοξοι με τα ίδια μας τα στοιχεία, ότι τα καθαρά κέρδη θα είναι πολύ μεγαλύτερα κατά πιθανότητα από το 1,5-2 δις που εμείς έχουμε εκτιμήσει για μια δεκαετή περίοδο μετά από την έναρξη των κεντροποιημένων υπηρεσιών. Τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία διαβουλεύσεων με τα 40 ε, κράτη-μέλη για να λάβουμε και τη δική τους έγκριση για τα επόμενα βήματα. Συζητούμε και με την Εκομισιόν για να δούμε τι είδου ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορούμε να λάβουμε για να αρχίσουμε ε, να έχουμε τα θετικά αυτά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν. Για να είμαστε σαφείς, έχουμε ζητήσει την σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών και να συνεχίσουμε τις κεντροποιημένες υπηρεσίες, αυτή την πρωτοβουλία μας, με την αξιοποίηση του προπολογισμού του Eurocontrol. Όμως έχουμε περιορισμένους πόρους και έχουμε και ε, το, ε, τους προεράτα στόχους μας, γι' αυτό και θα μας πάρει μερικά χρόνια ακόμα να πετύχουμε τους στόχους μας. Και αυτό βεβαίως δεν είναι η ιδανική κατάσταση. Θα θέλαμε λοιπόν και κάποια περαιτέρω στήριξη από το TNT. Ποια είναι τα ωφέλη από τη δική μας προσέγγιση. Μίλησα για την αποδοτικότητα και δεν μιλάμε μόνο για αποδοτικότητα σε ό,τι αφορά το κόστος, αλλά και τη λειτουργία, την αύξηση της ικανότητας και της ασφάλειας, τη βελτίωση της ασφάλειας. Όλα αυτά είναι θετικά, γιατί και οι στόχοι για τη δεύτερη περίοδο αναφορά ε, οριστικοποιούνται αυτή τη χρονική στιγμή. Τα ESPs ε, θα χρειαστούν τη βοήθειά μας ε, για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Και θεωρούμε ότι θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι σε εθνικό επίπεδο και μόνο. Οι κεντροποιημένες υπηρεσίες θεωρούμε ότι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κόστου των κατακαιρματισμένων υπηρεσιών. Ξέρω ότι στο ΣΕΣΑΡ και ιδιαίτερα οι αεροπορικές εταιρείε ε, ανυπομονούν να αρχίσουν τα θετικά αποτελέσματα μετά από τόσες, ε, τόσα χρόνια εξελίξεων. Οι κεντροποιημένες αυτές υπηρεσίες ε, θα μας βοηθήσουν να έχουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα αν εφαρμόσουμε τα προγράμματά μας με συνεκτικό τρόπο. Επιπλέον θα μας βοηθήσουν να διασφαλίσουμε ότι το ΣΕΖΑΡ και εν γέννη ο Ευρωπαϊκός ε, Ενιαίος Ουρανός ε, καλύπτουν ε, το σύνολο της Ευρώπης, κάτι το οποίο είναι σημαντικό αν θέλουμε να συνεχίσουμε τις βελτιώσεις που όλοι επιθυμούμε. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να καλύπτονται και τα 40 κράτη-μέλη του Eurocontrol. Και αυτό συνάδει και με την πολιτική γειτονίας της Ευρώπης αλλά και για την πολιτική σε ό,τι αφορά την ε, αεροπλοεία. Έχουμε και την ε, Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα τέτοια πρακτική που χρησιμοποιείται πλέον και από άλλε χώρε, όπω ε, ακόμα και η Νότια Αφρική ή η Νέα Ζηλανδία. Επομένω, εξάγουμε υψηλή τεχνολογία προ άλλα τμήματα του κόσμου και αυτό μπορεί να γίνει και με τι κεντροποιημένε υπηρεσίε, καθώ αποτελούν πραγματική δυνατότητα εξαγωγών ευρωπαϊκής ε, τεχνογνωσίας και υψηλής τεχνολογίας σε άλλα μέρη του κόσμου. Και έτσι θα έχουμε ανώτερη θέση στο παγκόσμιο προσκήνιο κατά το σχεδιασμό αυτών των υπηρεσιών. Σημαντικό είναι επίσης ε, όλο αυτό να πάει και στο, στο ICAO, στο Μοντρεάλ και μόνο έτσι μπορούμε να του πείσουμε ότι μπορούν να λάβουν υπόψη και τις δικές μας υπηρεσίες στον ΙΚΑΟ, στο Μοντρεάλ. Άλλο στοιχείο, η δημιουργία θέσεων εργασίας που είναι πάντα ένα λεπτό ζήτημα και πολύ χαίρομαι που ε, το φύγω εδώ, γιατί δεν θεωρούμε ότι οι κεντροπεμένες υπηρεσίες, αυτή η πρωτοβουλία θα ε, θέσει σε κίνδυνο θέσεις εργασίας, είτε στο Eurocontrol είτε στις εφιστάμενες ANSP. δεν σημαίνει ότι θα χαθούν ε, θέσει εργασία μόνο και μόνο επειδή πολλοί κόσμοι ασχολείται με τι κεντροποιημένε υπηρεσίε. Καθόλου. Κάποιε από τι κεντροποιημένε υπηρεσίε είναι νέε. Κάποιε έχουν ε, επεκταθεί στο πεδίο λειτουργία του και άλλε ε, υιοθετούν, θα αναλάβουν το ρόλο των ελεγκτών. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν και δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, γιατί δεν θα είναι το ίδιο το προσωπικό του Eurocontrol εδώ στις Βρυξέλλες που θα τρέχει το πρόγραμμα, είτε θα εμείς θεωρούμε ότι θα παραχωρήσουμε κάποιες από τις ε, δραστηριότητες που έχουμε αναλάβει και τις οποίες επιτελούμε αυτή τη στιγμή. Θα ζητήσουμε από τις NSP των ε, ευρωπαϊκών κρατών μελών να υποβάλουν προσφορά και να τρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε εθνικό επίπεδο. Μιλούμε και για τα 40 κράτη-μέλη του Eurocontrol. Και έτσι έχουμε και το άλλο όφελος ότι αυτές οι NSPs λειτουργούν και έξω από τα εθνικά του σύνορα, ε, ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ τους για την παροχή υπηρεσιών σε ε, πανευρωπαϊκό επίπεδο και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιες ANSPs. Εδώ θα πρέπει να πω όμως ότι κάποιες από αυτές δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κάποιες λιγότερο. Κάποιες ανησυχούν για το επίπεδο ελέγχου που θα έχουν σε ό,τι αφορά αυτές τις υπηρεσίες. Και εμεί ακριβώ θέλουμε να δούμε με αυτού του παρόχου υπηρεσιών πώ αυτό θα λειτουργήσει στην πράξη και τι μορφή θα πρέπει να λάβει η διακυβέρνηση. Όμως, εν γέννη, είχαμε θετικές αντιδράσεις και από τον τομέα της κατασκευής, ε, αλλά και από τις στρατιωτικές υπηρεσίες. Βεβαίως, οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείε είναι αυτές που ανυπομονούν περισσότερο, γιατί θεωρούν ότι οι υπηρεσίες ε, αυτές που θα είναι πιο συνεκτικές ε, και πιο οικονομικά αποδοτικές είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, που μπορεί να γίνει πιο σύντομα και με πιο συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως ανέφερα και στην αρχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξαιρετικά θετική. Πράγματι, το συμπεριέλαβαν αυτό το πρόγραμμα και στην πρόταση SES 2+. E θα το δείτε και στο ίδιο το κείμενο. Τώρα εγώ δεν θα επισέλθω σε αυτή τη συζήτηση για το SES 2+. E όμως ε, θα ήθελα να πω ότι αυτές οι κεντροποιημένες υπηρεσίες μπορούν και θα πρέπει να προωθηθούν αν θέλουμε οικονομικά αποδοτική ψηλή τεχνολογία να εφαρμόζεται στο μέλλον και με μείωση του κόστου. Οι κεντροποιημένε υπηρεσίε βεβαίω θα, μπορούσαν θα να θεωρηθεί μια μέση οδό μεταξύ του κατακαιρματισμού που βλέπουμε σήμερα και τη πλήρη αποσύνδεση των υπηρεσιών. Οι κεντροποιημένε υπηρεσίε, ε, κατά τη γνώμη μα, αποτελούν ε, μια ρεαλιστική συμβαστική λύση που μπορεί να επιτευχθεί και να εφαρμοστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά. Το SES 2 Plus επίσης προωθεί τον ρόλο του διαχειριστή δικτύου και είμαστε υπέρ. Είναι ένα ακόμα στοιχείο που θεωρούμε ότι είναι πολύ λογικό. Μάλιστα θεωρούμε ότι ο ρόλος του διαχειριστή δικτύου θα συνεχίσει να διευρύνεται γιατί έχει πραγματικό αντίκτυπο στην επίδοση του δικτύου, για παράδειγμα σε αφορά την αποφυγή καθυστερήσεων, τη μείωση των καθυστερήσεων και ε, την ε, χάρξη πιο ε, αποδοτικών πορείων έτσι με την εξοικονόμηση καυσίμων, εκπομπών και οικονομικών πόρων έγινε και μία μελέτη την οποία ζητήσαμε γιατί ε, ταυτοχρόνως αναθεωρούμε και τον ρόλο και τη δομή του Eurocontrol. Και κάθε οργανισμός θα πρέπει να ε, διερευνά κατά πόσο η λειτουργία του είναι κατάλληλη και μήπως θα πρέπει να βελτιωθεί. Έτσι, ερχόμαστε σε επαφή με τα διαφορετικά μέρη, ε, τα κράτη-μέλη και τις στρατιωτικές δομές ε, και τα αεροδρόμια και όλοι οι ενδιαφέρομενοι φορεί εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Θα συζητήσουμε ποια μορφή για κυβέρνηση είναι καλύτερη και κατά πόσο θα έπρεπε να εξετάσουμε μια ακόμα ευρύτερη συμμετοχή μελών. Για παράδειγμα, αυξανόμενο αριθμό πτήσεων ε, περίπτωση τη Ευρώπη. Κάτι το οποίο δεν βλέπαμε στο παρελθόν. Δεν είχαμε τέτοιε ε, πτήσει που περνούσαν πάνω από την Ευρώπη οι οποίες πλέον απευθύνονται και ε, κατευθύνονται μάλλον προς ε, τους, ε, τους μεγάλους κόμβους, αεροπορικούς κόμβους. Και γι' αυτό καλό θα ήταν να βελτιώσουμε τις συνδέσεις μας, ούτως ώστε το δίκτυό μας να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό και έτσι ο Eurocontrol να καταστεί ένας ακόμα πιο χρήσιμος εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτός είναι και ο δικός μας σκοπός, να είμαστε χρήσιμοι και να συνεργαζόμαστε μαζί με τα ενδιαφέρομενα μέρη, ούτως ώστε ο Ευρωπαϊκός ε, Ενιαίος Ουρανός να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φώστερ καταρχήν, καθώς ε, ήσασταν ε, οι μόνοι εδώ όταν ξεκινήσαμε. Τζάκι λοιπόν, μπορείς να επιτεθείς. Ευχαριστώ πολύ, πρέπει να φύγω πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ να μας συναντήσετε, κύριε Μπρένερ, από το Eurocontrol. Νομίζω ότι η χρονική συγκυρία είναι πάρα πολύ καλή, γιατί εξετάζουμε τον ενίο ουρανό 2 και φυσικά κάποια στιγμή ε, θα εξετάσουμε και την σχετική γνωμοδότηση. Η Κομισιόν ε, εργάζεται επίσης πάρα πολύ σκληρά έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να είναι πιο ενεργητικά σε αυτό το τομέα. Το δικό μου κρατος μέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ιδιαίτερα ενεργητικό και πιστεύει στα ωφέλη που θα προκύψουν από όλο αυτό και ο τρόπος που παρουσιάσατε τα επιχειρήματά σας και τα σχόλιά σας νομίζω ε, αντιμετωπίζει κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τις θέσεις εργασίας και την απώλεια θέσεων εργασίας γιατί οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι αυτά θα ισχύουν ε, όσο προχωρά ο χρόνος. Υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο περιοδικό Flight ε, αυτή την εβδομάδα και βέβαια θα υπάρχει και ανταγωνισμός με το Σέσαρ και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ήδη κάνουν δοκιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, ε, θα είναι πολύ σημαντικό και για το ποσό της τεχνολογίας που θα θέλουμε, το ποσό της τεχνολογίας που θα θέλουμε να πωλήσουμε. Εκ μέρους, ε, λοιπόν, ε, του ECR σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Έχετε υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Μαρινέσκου, εισηγητής, βρίσκεται και εδώ σήμερα και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε να προχωρήσει το θέμα, γιατί τα ωφέλη που παρουσιάσατε σχετικά με τα καύσιμα για το θέμα του ανταγωνισμού, της τιμολόγησης, για όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να τα αγνοήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι από το ECR και ανυπομονώ να σας ξαναδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προφορική παρουσίαση. Έχω μόνο κάποιες γρήγορες ερωτήσεις για τις συγκεντρωμένες υπηρεσίες. Είπατε ότι υπάρχουν πάροχοι υπηρεσιών που συμφωνούν με αυτό και άλλοι που διαφωνούν. Ξέρω ότι γενικά συμφωνούν επί τη αρχής, αλλά δεν συμφωνούν με όλες τις υπηρεσίες. Επομένως, υπάρχει μια διαίρεση σε δύο ομάδες, ε, δηλαδή κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το διορθώσετε. Είπατε κάτι σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του κόστους. Πρέπει να συζητήσετε μαζί τους. Γιατί τα όσα λένε δεν βασίζονται σε κάποια ανάλυση κόστους ωφέλους. Δεύτερον, αναφερθήκατε στο θέμα του διευθυντή και είπατε ότι είστε ικανοποιημένος που θα έχει ένα μεγαλύτερο ρόλο να ασκήσει στο σες ΣΥΝ. Τι πιστεύετε σε σχέση με το διαχωρισμό του διευθυντή, του δικτύου, ε, δηλαδή να καταστεί ένας ανεξάρτητος φορέας από το Eurocontrol και τι γίνεται με το PRB Δεν γίνει η οικονομική ρυθμιστική αρχή, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι λογικό να είναι ανεξάρτητος φορέας από το Eurocontrol. Τι πιστεύετε για όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριος Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρένα για την παρουσίαση. Τόσο ωραία που δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι και αληθινά. Σαν να έχουμε κερδίσει το πρώτο λαχείο. Άρα και τα κράτη-μέλη μπορούν να κερδίσουν πολλά λεφτά με τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες και αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της ασφάλειας των πτήσεων γιατί είναι βέβαια θέμα ε, που αφορά όλα τα κράτη-μέλη το να υπάρχει επαρκής ε, διασφάλιση των πτήσεων. Η ασφάλεια λοιπόν είναι πολύ σημαντική και αυτή. Και έχω με δύο ερωτήσεις. Μια και είπατε ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να αναθέσουν στις αρμόδιες ε, για την ασφάλεια αρχές νέα καθήκοντα με κεντρική βέβαια οργάνωση ε, μέσω της ΙΑΤΑ και της Eurocontrol έστω. Αλλά συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη με αυτήν την κατανομή των αρμοδιοτήτων και με ποια κριτήρια γίνεται αυτή η κατανομή. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε, αν δηλαδή γίνεται η κατανομή σωστά και βέβαια αν τελικά ο τελικός αποδέκτης της Επίσης, θέσεις εργασίας. Εάν καθούν θέσει εργασία, δεν ε, δημιουργούνται νέε, εξάγεται αυτή η ψηλή τεχνολογία. Σε αυτές τις κεντροποιημένες λοιπόν κεντρικά οργανωμένες υπηρεσίες θα υπάρχει αποκέντρωση ως προσορισμένες αρμοδιότητες οι οποίες ενδεχομένως θα ανατεθούν σε τοπικές αρχές ασφαλείας των πτήσεων και ποιες θα είναι αυτές. Τελευταία ερώτηση. Με αυτές τις προτάσεις σας, η Eurocontrol γίνεται πιο φθηνή για το κράτη-μέλη. Γιατί από ό,τι ακούμε η Eurocontrol έχει πάρα πολλούς υπαλλήλου και μάλλον δεν είναι και τόσο αποτελεσματική από ό,τι λένε οι επικριτές σας τουλάχιστον. Ευχαριστώ Κράμερ. Ναι, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω για την παρουσίαση. Στο τασταπεινά, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που δεν ήμουν παρόν στην αρχή της συνεδρίασης. Δύο όμως πολύ σημαντικοί προσκεκλημένοι μου ήταν, ε, με απασχόλησαν στην αρχή της συνεδρίασης, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται εδώ τώρα για να συμμετάσχουν στη συζήτησή μας. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τις προτάσεις. Η συζήτηση έχει ήδη γίνει εδώ για τους ευρωπαϊκούς εθέρες. Είναι όλα αυτά ξεκάθαρα, είναι ήδη ρυθμισμένα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, απλώς τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να παραβιάζουν τη διαδικασία. Τι θα κάνετε λοιπόν για να πείσετε τα κράτη-μέλη να, να σεβαστούν την νομοθεσία και πώς μπορείτε να τα πείσετε και τι είδους απαντήσεις σας προσφέρουν όταν ε, ε, τα φέρετε ενώπιον των ευθυνών τους. Ο κύριος Κόχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρένερ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Χρόνια τώρα ασχολούμαστε με τους νέους ευρωπαϊκούς ουρανούς και έχετε τώρα με την ε, πρόταση αυτή για τις ε, κεντρικά οργανωμένες ε, υπηρεσίες την ευκαιρία να προχωρήσετε. Βλέπω κάποια πλεονεκτήματα, αλλά ήθελα να μου πείτε στα προβλήματα που εντοπίζονται πέραν των πλεονεκτημάτων, πού εντοπίζετε εσείς λόγους δυσκολιών, πού είναι τα προσκόμματα. για τον έλεγχο τώρα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πολύ πιο αποτελεσματικέ από ότι Ευρώπη στο θέμα του ελέγχου και τη ασφάλεια. Θα μπορέσουμε με του ε, νέου ευρωπαϊκού ευθέρε να το καταφέρουμε αυτό, ή χρειάζεται ένα άλλο πλαίσιο. Ευχαριστώ. Άλλο κανεί θέλει το λόγο πριν να μιλήσω κι εγώ. Οι ερωτήσει που ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν ε, κάποια πράγματα που το υπόθηκαν. Δηλαδή, πώ θα πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι αυτό είναι ο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί πραγματικά δυσκολευόμαστε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν το οτιδήποτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία. Και κάποιοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσουν τα κράτη-μέλη όταν μιλάμε για το θέμα των μεταφορών, αλλά ιδιαίτερα δυσκολευόμαστε στο θέμα τη ε, διαχείριση των ενέργειων μεταφορών και νομίζω ότι με επιτυχία καταφέρατε να αποφύγετε να αναφέρετε τον ενιαίο ουρανό, τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ουρανό 2+. Συν, ε, ξέρω κάποιοι κάποια κράτη-μέλη καλούν για ε, απόρριψη του ΣΕΣ 2+, κυρίως σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό των υπηρεσιών. Και τα εις δύο τελευταίες εβδομάδες γίνει φιάλτη σε αυτήν την Επιτροπή το θέμα του ε, διαχωρισμού. Και επίση αναφερθήκατε και στην απώλεια θέσεων εργασία Είναι ενδιαφέρουσα η ανάλυση αυτή γιατί τα συνδικάτα είναι απολύτως πεπισμένα ότι θα υπάρχουν απολύσεις, τις συνεργασίες και επομένως έχουμε αυτό το πρόβλημα της αντίληψης. Δηλαδή εσείς λέτε όχι, δεν θα υπάρχουν απώλειες στις συνεργασίες, θα υπάρχουν περισσότερες στις συνεργασίες, αλλά υπάρχει μια αντίληψη και έξω ότι θα υπάρξει απώλεια συνεργασίες και ότι ε, είδαμε ότι πριν δύο εβδομάδες είχαμε κάποιες διαμαρτυρίες εδώ στην πλατεία και το ίδιο θα ξαναγίνει. Και πώς ε, λοιπόν θα αλλάξουμε την αντίληψη που υπάρχει στον κόσμο ότι όλα αυτά το σες το ΣΕΣ2, το ΣΕΖΑΡ δεν θα οδηγήσουν σε πολύ θέση Κύριε Μπρένερ, ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μπλοκ. Η μία ερώτηση αφορούσε τι συγκεντρωμένε υπηρεσίε, τι εννέα συγκεντρωμένε υπηρεσίε. Εγώ είπα ότι αυτέ οι εννέα υπηρεσίε που έχουμε εντοπίσει όλε έχουν να κάνουν με τα δεδομένα, δεν ε, μιλάμε για συγκεντρωμένες υπηρεσίες ε, διαχείρισης της ενέργειας κυκλοφορίας, αλλά μιλάμε για συγκέντρωση της παροχής των δεδομένων ε, σε τόπους όπου έχει λειτουργήσει ο έλεγχος. Τώρα η τεχνολογία που αναπτύσσεται στο ΣΕΣΑΡ επιτρέπει να μην χρειάζεται επεξεργασία όλα τα δεδομένα, αλλά να έχουμε επεξεργασία σε ένα κεντρικό περιφερειακό επίπεδο και κατόπιν να διατίθεται στα κέντρα διαχείρισης του ενέργειας κυκλοφορίας. Δεν έχει σημασία λοιπόν από πού προέρχονται αυτά τα δεδομένα, είτε από το σελίδι, από μια κεντρική τοποθεσία. Εμείς ε, θέλουμε να έχουμε δεδομένα υψηλής ποιότητας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα, οι υπηρεσίες ε, που δίνουμε είναι έξι υπηρεσίες, όχι σε μία πλήρη μορφή. Και εδώ ε, έρχεται η Eurocontrol, δεν θέλει να πάρει τίποτα από τους ΕΕΝΕΣ πίσω από τους παρόχους υπηρεσιών αεροπλοείας. Εδώ έχουμε προτείνει έξι υπηρεσίες που προέρχονται από εμά και έχουν να κάνουν με το συνδεσμό της συχνότητας. Δεν υπάρχει λοιπόν επικάλυψη. Ε, με τα αεροσκάφη, με τα μηνύματα που στέλνονται με πληροφορίες και κτλ. Αυτές είναι, αυτά είναι έξι σύνολα υπηρεσιών που παρέχουμε σήμερα και θέλουμε να τα επεκτείνουμε. Δύο από τις εννέα υπηρεσίες σήμερα παρέχονται από τους παροχούς υπηρεσιών αεροπλοείας και έχει νόημα να παρέχονται σε πιο κεντρική βάση και η ένατη υπηρεσία είναι μια συνδυασμένη υπηρεσία μεταξύ των ANSP, των παροχών υπηρεσιών και της Eurocontrol. Έτσι λοιπόν φέρνουμε το μεγαλύτερο πακέτο των υπηρεσιών ε, στη Eurocontrol και οι υπαροχοι υπηρεσιών κατανοούν ότι κάτι συμβαίνει και μάλιστα συνεισφέρουμε τα συνδικάτα της Eurocontrol έχουν συνεργαστεί στενά μαζί, σας, μαζί μας και μπορώ να σας πω ότι όταν πρωτοδημιουργήσαμε την πρόταση αυτή δεν ήταν και ιδιαίτερα ενθουσιασμένα αλλά το δέχτηκαν και είπαν ότι αν τελικά δεν προχωρήσουμε και δεν υποστηρίξουμε και κάποιες από τις δικές μας υπηρεσίες τίποτα δεν θα προχωρήσει έτσι λοιπόν δεν ε, θέλουμε να φύγουν αυτές οι υπηρεσίες αλλά το υποστηρίζουμε και συνολικά έχουμε να υποστηρίξουμε, έχουμε ρόλο να παίξουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν συνέβη σε σχέση με το Eurocontrol και τα συνδικάτα. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριο Μαρινέσκου, ναι, κάποιοι υπάρχουν υπηρεσιών πιστεύουν ότι δεν ήταν καλό να πάρουν αυτέ τι έξι υπηρεσίε της Eurocontrol ως τμήμα του πακέτου που προτείνονται στη δική του ε, αρμοδιότητα και να μην συνεισφέρουν με τι ε, δύο που έχουμε προσδιορίσει. Εμεί ε, θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση και να εργαστούμε λεπτομερώ για το θέμα του εφικτού, δηλαδή αν έχουν νόημα αυτέ οι δύο υπηρεσίε το εφικτό δεν σημαίνει η σκοπιμότητα, δεν ε, σημαίνει ότι έχει ε, ληφθεί ήδη μια απόφαση, αλλά νομίζω πρέπει να υπάρχει βούληση να συνεργαστούμε και να διερευνήσουμε εις βάθος τι συμβαίνει με αυτές τις δύο υπηρεσίε. Και κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες έχουν να κάνουν με τα δεδομένα ραντάρ και δεν υπάρχει συνεκτικότητα στην Ευρώπη, γι' αυτό η Eurocontrol προτείνει μια κεντρική διάθεση αυτών των δεδομένων. Τώρα, σε σχέση με το CBA, όταν ξεκινήσαμε το δικό μας πακέτο, φτάσαμε στα 150-200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και ε, το πολλαπλασιάζουμε αυτό με 10 χρόνια. Φυσικά μας ρώτησαν μπορείτε να αξιολογήσετε, μπορεί κάποιος ανεξάρτητος οργανισμός να αξιολογήσει αν ισχύουν αυτά τα νούμερα. Τα κράτη-μέλη έθεσαν αυτή την ερώτηση και προσέλαβαν μια εταιρεία και τελικά το πόρισμα ήταν ότι είναι πολύ συντηρητικά αυτά τα δεδομένα και εγώ ήθελα να έχω πολύ συντηρητικά δεδομένα γιατί αυτό δεν ήταν ένα ε, επιχείρημα προς, ε, για την πώληση. Είναι κάτι σημαντικό, είναι μία συνεισφορά, αλλά περισσότερο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το μοντέλο που κρύβεται από πίσω και όχι τόσο το αριθμητικό στήριο. Αυτό δεν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητά υψηλά νούμερα για να πείσουμε, αλλά θέλαμε καλύτερα συντηρητικά νούμερα. Η εταιρεία που επιλέχθη, που εξέτασε τα νούμερα, είπε είναι αξιόπιστα αυτά τα δεδομένα και είναι συντηρητικά. Κατόπιν ήρθαν ε, τα κρατημέλη και τα 39 και είπαν ε, τώρα θα ε, βάλουμε και εμείς τους δικού μας οικονομικούς εμπειρογνώμονες να αξιολογήσουν τι έχει κάνει η Eurocontrol. Αυτό ήταν το τρίτο βήμα. Είχαμε την Επιτροπή των Κρατών Μελών για τα χρηματοοικονομικά και τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υποστηρίζει αυτά τα αριθμητικά στοιχεία και ότι είναι αξιόπιστα ακόμη και αν είναι συντηρητικά τώρα. Ε, οι παρόχοι υπηρεσιών ε, δεν ε, μπορούσαν να λάβουν όλα τα στοιχεία που πήραν τα κράτη-μέλη και εδώ υπάρχει ένας λόγος γιατί αν ζητήσει κάποιο ένα διαγωνισμό από τους παρόχους υπηρεσιών να παρουσιάσουν προσφορά για αυτές τις υπηρεσίες και έχεις βάλει επιτάπητος, έχεις αποκαλύψει τα νούμερα, ήδη ξέρουν αυτοί ποιο είναι το αποτέλεσμα. τα κράτη-μέλη πήραν τα στοιχεία αυτά μέχρι το τελευταίο ψηφίο και κατέληξαν στο συμπέρασμα σε σχέση με το αν ε, είναι πιο ακριβή γεροκοντρόλο, Όχι, περάσαμε δύσκολου καιρού. Τα τελευταία πέντε χρόνια μειώσαμε το προσωπικό από 2.500 σε 2.000. Δεν ήταν εύκολη αυτή η διαδικασία και σα διαβεβαιώ, ήταν πάρα πολύ δύσκολη παρόλα αυτά, αυτή ήταν η προπαρασκευαστική δουλειά μας για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στους στόχους επίδοσης. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή λέμε έχουμε δεσμευτεί πλήρως για να μειώσουμε τα τέλη χρήσης και εμείς συμβάλλουμε στο να πετύχουμε τους στόχους επίδοσης. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να είναι προϋπόθεση κατάθεσης μια τέτοιας πρότασης. Η ιδέα αυτή δεν έρχεται από την πίσω για να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες ή περισσότερα χρήματα, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη να προχωρήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, πιστεύουμε ότι αυτό που υπάρχει είναι κάτι πολύ καλό. Έχετε όλους τους πάροχους εκεί, έχετε και τα αεροδρόμια και το στρατιωτικό σκέλος και τις χρήστε. τους ε, γιατί λοιπόν να μην επεκτείνουμε αυτό το δίκτυο έτσι ώστε να έχουμε και ένα πακέτο συγκεντρωμένων υπηρεσιών. Τα κράτη-μέλη το υποστηρίζουν, λένε ναι, θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα ατόμων που θα προβαίνει στη διακυβέρνηση, η Eurocontrol και ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να είναι διευθυντές του προγράμματος. Αυτή είναι η πρότασή Έτσι λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε τον κανονισμό του Διευθυντή για να καλύπτει και αυτή τη διακυβέρνηση που γίνεται βάση του κλάδου. Τώρα για το ERB, αν θα έπρεπε να είναι εντό ή εκτό ε, τη αρμοδιότητα Eurocontrol. Η Eurocontrol έχει με ένα συμβόλαιο με την Κομισιόν που υποστηρίζει τι δραστηριότητε του PRB. Δεν ε, επηρεάζουμε τι δραστηριότητε του PRB ε, αυτού του συμβολίου καθόλου ε, γιατί τα μέλη του εκλέγονται ανεξάρτητα και δεν έχουμε λόγο εμείς για το ποιος εκλέγεται. Εμείς τι κάνουμε διαθέτουμε τα δεδομένα που θέλει το Συμβούλιο και κάνουμε μία ανάλυση. Οποιαδήποτε ανάλυση μας ζητήσει το Συμβούλιο, δίνουμε τα στοιχεία, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις. Όμως αυτό που κάνουμε είναι ότι τα δεδομένα αυτά τα στέλνουμε και στο PRC που είναι μια ομάδα της Eurocontrol που έχει να κάνει, που καλύπτει όλα τα μέλη και τα 40 μέλη της Eurocontrol, όχι μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να πάνε προς μία κατεύθυνση μέτρησης, αν πάνε προς μία τέτοια κατεύθυνση μέτρησης που δεν θα συνάδει με το PRB, τότε καλό είναι να υποστηρίζουμε την ε, PRC. Έτσι λοιπόν η αφαίρεση από το Eurocontrol θα έθετε το ερώτημα ποιος ε, κάνει την υποστέριξη. Το, ε, τι θα γίνει όταν ε, οι δύο ομάδες θα πήγαιναν σε αντίθετες κατευθύνσεις αν δεν υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ των δύο ομάδων και αν δεν συμμετέχουν και τα δύο άτομα στα δύο αυτά συμβούλια, που αυτή τη στιγμή είναι ένα συμβούλιο. Αυτή είναι η ανησυχία μου, δηλαδή να μην υπάρχει περαιτέρω κατακαιρματισμός, αλλά σε ό,τι αφορά την μεγαλύτερη ανεξαρτησία, η Eurocontrol δεν ε, επηρεάζει σε καμία περίπτωση το Συμβούλιο, το PRP, δεν εκλέγονται οι άνθρωποι από τη Eurocontrol. Σε σχέση με το τι λένε τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη, καθώς και συμμετείχα και στη συνδιάσκεψη στο Βίλνιους, είπαν ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα με το ΣΕΣ συν, αλλά είπαμε με συντριπτική πλειοψηφία επίση ότι είμαστε έτοιμοι να έχουμε μια περιορισμένη αγορά ε, για τις υπηρεσίες υποστήριξης ε, του ENSP. Έτσι λοιπόν, αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τα κράτη-μέλη το Δεκέμβριο και ελπίζω να θυμούνται τι είπα στο Βελίνους και να μην το ξέχασαν. Θα δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί αυτό. Γεια. Yeah το θέμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Ναι, ω Eurocontrol έχουμε ένα εργαλείο σύγκριση με τις ΗΠΑ. Αυτό γίνεται από ε, το Φορέα αναθεώρηση των Επιδεώσεων. Ο Eurocontrol υποστηρίζει αυτή την ε, δραστηριότητα. Πράγματι, οι ΗΠΑ παρέχουν ε, την ίδια ποιότητα και για μικρότερο κόστος, 40-50% μικρότερο κόστος από αυτό που χρεώνουμε στην Ευρώπη. Γιατί, γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα σύστημα, ενώ εμείς έχουμε 28 ή ακόμη και 40 πάροχους υπηρεσιών, έχουμε διαφορετικές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους ε, και, αν δεν, και δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη στιγμή τις συνθήκες εργασίας ε, και τον ε, το θεσμικό πλαίσιο, ε, μπορώ να σας πω ότι αν θέλουμε να είμαστε αντιγωνιστικοί πρέπει να βρούμε ένα αντιστάθμισμα και μόνο στο μέσο που βρήκαμε είναι να αναπτύξουμε υψηλές τεχνολογίες που δεν έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες που μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή σε μια κεντρική περιφερειακή βάση που θα προέρχονται από το ΣΕΣΕΡ και θα μειωθεί σημαντικά το κόστος και αυτό κάναμε με την πρόταση και είμαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει και η βάση δεδομένου IAS θα, θα, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Ταϊλάνδη, την Νότια Αφρική. Νομίζουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και εμεί αυτό. Τώρα η ερώτηση ήταν πώ να επεκτείνουμε αυτέ τι υπηρεσίε, γιατί πάροχοι υπηρεσιών εργάζονται σε εθνική βάση. Υπάρχουν πολλοί πάροχοι υπηρεσιών που θα ήθελαν ε, να επεκταθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα, αλλά δεν μπορούν γιατί υπάρχει εκεί ένα άλλο πάροχο υπηρεσιών που παρέχει το πλήρε σύνολο των ε, υπηρεσιών ε, και αν ε, τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίξει την ιδέα να χρησιμοποιηθεί μια πολύ μικρή αγορά υποστήριξης ε, της διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας, ε, τότε τελικά μπορούμε να έχουμε έναν πάροχο που θα παρέχει την υπηρεσία σε ευρωπαϊκή βάση. Πρέπει να θέσουμε κριτήρια έτσι ώστε να έχουμε μια κάλυψη και των κρατών μελών που δεν ανήκουν, κρατών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε παροχή αυτών των υπηρεσιών και αποδοχή των υπηρεσιών πέρα από τους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με συγχωρείτε αν ε, ξέχασα κάτι Α, για την απολύθεση συνεργασίας. Ε, τι κάνουμε. Φυσικά, οι κεντρικές υπηρεσίες έχουν πάντοτε την τάση ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι απόλυτα θέση, να υπάρχει απόλυτα θέση συνεργασία. Όμως γιατί δεν υπάρχει κάποια τέτοια προπτική στις υπηρεσίες που προτείνουμε, γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει παραδείγματα που, όπου δεν πέφτουμε κατευθείαν πάνω στο πρόβλημα των απολύσεων στις ενέπηρεσίε που προτείναμε. Έχει γίνει και μελέτη αντικτύπου και το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη συνεργασία. Τώρα, αν υπάρχει γενικό διαχωρισμό, τότε μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και μπορεί εκεί να έχουμε απόλυτη εργασία. Όμως για αυτές τις υπηρεσίες η υπόσχεσή μας είναι ότι δεν έχουμε θέμα τη συνεργασίας γιατί ε, δεν θέλουμε να τορπιλήσουμε τη δική μας ε, πρόταση και γι' αυτό επιλέξαμε αυτές τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ κύριε Πρένερ για την έκθεση. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Ασφαλώς θα σας ξαναθούμε όχι μόνο στην τρέχουσα, αλλά και στην προσεχή θητεία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε και καλή τύχη σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Ξέρετε ασφαλώ ότι εμείς εδώ σε αυτήν την Επιτροπή δεν τρέφουμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Γιατί συνήθω αυτά που υπόσχονται δεν τα τηρούν. Αν τα καταφέρετε εσεί, θα είστε ο πρώτος. Και πιο ικανό ασφαλώς από ότι εμεί. Σα ευχαριστώ θερμά. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε πρόσωπα εδώ στο Προεδρείο. So, next item is to carry on the... Το επόμενο θέμα είναι οι εκθέσεις των συντονιστών TNT. Σας προσπαθήσουμε να επιδείξουμε λίγη πειθαρχία γιατί χτες απαιτήχαμε παταγωδός. Παρακαλώ λοιπόν τους συντονιστές να μην περιοριστούν στα 7 λεπτά για τις παρουσιάσεις. Πρώτος ο Πέτερ Βάλας. Παρίσι Στρασβούργο. Έργο 17. Παρίσι Στρασβούργο, Στουτχάρβε. Βιέννη, Μπρατισλάβα. Πίτερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή σας ότι το έργο 17 Παρίσι Μπρατισλάβα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις περισσότερα, στα περισσότερα τμήματα έχουμε 600 χιλιόμετρα, περίπου τα μισά καλύψει με αναβάθμιση της γραμμής σε σχέση με την αρχική φάση του 2005. Για 450 χιλιόμετρα συνεχίζονται τα έργα και έχουμε 200 χιλιόμετρα όπου οι υπηρεσίε προσφέρονται με παραμέτρου τη προηγούμενη περίοδου. Θα σα δώσω μερικά παραδείγματα. Στη Γαλλία, η σύραγγα που διασχίζει τη Σαβέρνη προχώρησε σημαντικά για να ολοκληρώσει τον Πέντρο Κουρ Βέρντενχάιμ. Στη Γερμανία έχουμε βελτίωση σημαντικών ε, διασυνδέσεων για το αεροδρόμιο του Μονάχου το Neuen Kurve, το BILPA, το Financing και έτσι βελτιώνεται η διασύνδεση προσφορά μέχρι το 2018 θα έχει ολοκληρωθεί ε, προς Ανατολάς Μίλντορφ Σάλσπουργκ. Και εδώ έχουμε αρκετά παραδείγματα. Αλλά κυρίως Βιέννη Σάνκτ Πέλτεν με επιτάχυνση των επικοινωνιών και μείωση κατά 17 λεπτά του χρόνου της εδρομής, η σύραγγα του Λάιντσελ και η αναβάθμιση του κεντρικού σταθμού της Βιέννης έχουν προχωρήσει επίσης. Προβλήματα υπάρχουν Η αύξηση του κόσμου, παραδείγματι, για την, περίο για την ε, διαδρομή Βέλτλιγκερ-Ούλμ. Προβλήματα σχετικά με τη Στουτχάρδη η Σλοβακία επίσης η σχεδιαζόμενη βελτίωση από τη Βιέννη μέχρι την Πρατισλάβα ε, με κάποιες καθυστερήσεις που όμως υποσχέθηκε ο Υπουργός των Μεταφορών της Σλοβακίας ότι θα αντιμετωπίσει ταχαίως. Ε, κύριε Πρόεδρε, το φυλάδιο που βλέπετε είναι κατά πιθανότητα και η τελευταία έκθεση που θα υποβάλω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έργο προτεραιότητας υπαριθμών 17, γιατί ολοκληρώνεται εδώ η θητεία μου σιγά σιγά. Το 2005 επιμελούμε με μια μικρή διακοπή των, των θεμάτων. Έχω συλλέξει μπορώ να πω μια κάποια εμπειρία σχέση με το συντονισμό του έργου. Πολύ ευχαριστώ να τη μοιραστώ μαζί σας. Στο χρόνο που έχουμε στη θέση μας φυσικά. Και αυτό σημαίνει ότι θα κάνω πολύ σύντομε παρατηρήσει, λίγε παρατηρήσει. Είναι σημαντικό τέτοια project, τέτοια έργα να προχωρούν πέραν των εθνικών συνόρων, πέραν του ε, σιδηροδρόμου, δηλαδή διαλειτουργικότητα και πέραν της μίας και μόνο γραμμή, δηλαδή ανάπτυξη πολλαπλών διασυνδέσεων. Θα ήθελα ιδιαίτερα να επίσης την προσοχή όλων των συναδελφών και του Κοινοβουλίου εν γέννη ως προς μία από τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε διαρκώς. Ούτε για ένα λεπτό δεν μπορούμε να λησμονήσουμε την ανάγκη να εξασφαλίζεται η υποστήριξη της κοινή γνώμη. Πρέπει πάντα να επανερχόμαστε στην κοινή γνώμη, να εξηγούμε, να αναπτύσσουμε ανταλλαγή απόψεων με τους πολίτες και επίσης αλλάζουν ταχύτατα κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη, αλλά και οι τοπικές κυβερνήσεις. Και μπορεί τα προβλήματα να είμαστε σε θέση ε, να τα αντιμετωπίσουμε όσον αφορά το κοινό, την κοινή γνώμη. Έχω δει από ενώσεις και συνδέσμους πολιτών, με κυβερνητικές οργανώσεις, όπως ε, ο Σύλλογος ΤΣΒ Ανατολάς, η Μαγκιστράλα Ευρώπα, ε, που με έχουν υποστηρίξει τα μάλα για δε τις ταχείες φυσιολογικές και συνήθεις αλλαγές κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη, τα θεσμικά όργανα, η πρώτο, πρώτο το Κοινοβούλιο, αλλά και ε, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μου έχουν προσφέρει πολύ σημαντική βοήθεια. Καλό λοιπόν και το προσεχές, την προσεχή θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας στηρίξει, γιατί τώρα περνάμε σε πολύ δύσκολο σχεδιασμό, σχεδιασμό υψηλού επίπεδου για την πολυτροπικότητα. Αν δεν μπορέσουμε λοιπόν να πείσουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν μία γραμμή και ένα μόνο σιδηρόδρομο, μία μόνο σιδηροδρομική γραμμή, φαντάζεστε πόσο δύσκολο θα είναι να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη αλλά και τη χρηματοδότηση των κρατών μαλλών για την πολυτροπικότητα με τα περιορισμένα κονδύλια που έχουμε στο, πλαίσιο, στο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε δηλαδή και νόμιμο αίρισμα αλλά και πολιτική ε, υποστήριξη. Ευχαριστούμε πολύ Πίτερ. Ευχαριστώ που δεν μακρηγόρησες κιόλα. Έμεινε στο χρονικό όριο. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Κράμερ, Μάισνερ. Άλλος κανείς. Γκουμάια. Μάλλον δεν είναι τυχαίο που ήταν ο μόνος που κατάφερε να μείνει στο χρονικό του όριο, γιατί δεν είναι μόνο εξαίρετος καθηγητής ε, πανεπιστημίου στην Ουγγαρία, αλλά ήταν και υπουργό ε, εξωτερικών. Υπήρξε και επίτροπος, όμως σίγουρα ξέρει πως ε, πρέπει κανείς να τηρεί τα χρονικά όρια. Χαίρομαι ιδιαίτερως ε, που εκπονείστε ένα τέτοιο ε, έργο. Ελπίζω να είστε και ε, υπουργό Εξωτερικών και πάλι στο μέλλον στην Ουγγαρία. Να μην... Να αλλάξετε και πάλι λοιπόν πεδίο. Είναι σημαντικό αυτό το πεδίο λοιπόν για μα. Όμω πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει μια καλή σύνδεση με την Πρωτεσλάβα για την Βουδαπέστη. Είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Είναι εξαιρετική ομάδα σας. σε όλη την εισαγωγή και στη σύνοψη έχετε παρουσιάσει τα όσα κάνατε. Το δικό μου ερώτημα είναι ποιες συμβουλές μπορείτε να δώσετε στον στον ε, διάδοχό σας, ε, πώς ε, μπορεί να συνεχίσει η επόμενη ομάδα. Και τώρα βεβαίω βρισκόμαστε εν μέσω κρίση και η κρίση πάντα αποτελεί μια πρόκληση για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά μια κατάσταση. Ποια είναι η δική σας γνώμη λοιπόν από την επαγγελματική σας πείρα σε ό,τι αφορά το ε, έργο προτεραιότητας ε, υπαριθμών 17. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το έργο σας. Ξέρετε ότι στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία πολλά θα αλλάξουν, πάρα πολλά μέλη θα αλλάξουν, επομένως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια καλή Επιτροπή Μεταφορών. Κύριος Κράμερ, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Χρόνια τώρα εργαζόμαστε κύριε Μπάλλας μαζί. Συγκεκριμένες ερωτήσει έχω. Έχω πολλές φορές διερωτηθεί για τον ε, σταθμό της Τουτχάρδης και έχω ρωτήσει αν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς μου απαντάτε πάντα ότι είναι εθνικό έργο, τοπικό έργο, δεν χρηματοδοτείται, όμως βλέπω ότι ε, σας ε, αμφισβητούν οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί φαίνεται ότι κάποια κονδύλια έχουν πάει στο σταθμό αυτό της Τουτχάρδης, ο οποίος μάλιστα είναι πολύ κατώτερος ως προς το δυναμικό του από τον υφιστάμενο είναι δε και σε κεκλειμένο επίπεδο και ως εκ τούτου δεν, είναι καθόλου, δεν εγγράφεται στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και δεν καταλαβαίνω τι έχει χρηματοδοτηθεί. Χρειάστηκε βέβαια πολλές φορές να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μου απαντήσει ότι από το Βέντρικερ μέχρι το ε, Ούλμ η γραμμή κόστισε 3 δις, το διπλάσιο πότε αρχικά είχε ε, σχεδιαστεί και ότι έχουμε μία διαμόρφωση του κόστου αυτού, ε, όπως και για το Κάισλιγκερ που όμως τελικά δεν ε, χρησιμοποιείται, όπως για το Παρίσι-Μπρατισλάβα που τελικά προσαρμόζεται για να μπορέσει να σηκώσει και φορτίο η γραμμή αυτή. Επειδή η Στουτχάρδη θα έχει μόνο επιβάτες, τότε μένει μόνο η γραμμή Παρίσι-Μπρατισλάβα ως μόνη για ε, που μπορεί να σηκώσει εμπορεύματα, ε, μεταφορά φορτίων δηλαδή, ε, αλλά τελικά νομίζω ότι αυτό στην πραγματικότητα δεν θα ισχύσει. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε για το αντίθετο. Και έχω πολλές φορές ρωτήσει και θέλω να το ξαναδούμε. Έχει γίνει μια συζήτηση για το ποια γραμμή περνάει από Βιέννη για Πρατισλάβα μέσω αεροδρομίου Βιέννης ε, προβλέπετε λοιπόν όντως να τεθεί σε λειτουργία αυτή η γραμμή βγαίνει αεροδρόμιο, Μπρατισλάβα με τη στάση του αεροδρόμιο που είχε, πολύ, είχε προξενήσει πολλές ε, αντιρρήσεις. Κυρία Μάισνερ, πρόεδρε ευχαριστώ. Κύριε Μπάλας και σε εσάς. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε. Σύντομες οι δικές μου ερωτήσεις, φαντάζομαι και πιο εύκολο να απαντηθούν είπαμε στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη να μην βλέπουμε μόνο εργοτάξια αλλά και ολοκληρωμένα έργα. Μέχρι το 2020 το αργότερο πρέπει να είναι ολοκληρωμένα όλα αυτά. Ε, ίσως να μην είναι εύκολη απάντηση τελικά, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να τηρηθεί αυτό το χρονικό όριο. Στις δε υπερσυνοριακές ε, διασυνδέσεις, οποίες έχουμε δώσει την προσοχή, προσοχή μας ιδιαίτερα, καθώς τα κράτη-μέλη δεν είναι τεθειμένα να τις χρηματοδοτήσουν το καθένα χωριστά, στο Στρασβούργο και στη γραμμή του Στρασβούργου και στη γραμμή της Μπρατισλάβα, η διασύνδεση με την ε, Μπρατισλάβα, φαίνεται ότι έχουν προσφέρει τα κράτη-μέλη επαρκή χρηματοδότηση. Και άρα δεν θα αποτύχει αυτό το έργο λόγω προβλήματος χρημάτων. Είναι αλήθεια αυτό. Κύριε Μπάλας. Αν μου επιτρέπετε. Θα ξεκινήσω με τις ε, τελευταίες δύο ερωτήσεις ή σειρά ερωτήσεων, σειρές ερωτήσεων. Καταρχάς για τον σταθμό Στουτχάρδης. Οι συντονιστές ετυπώνουν προτάσεις. Τις αποφάσεις τις λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη. Και πιστεύω ότι εν τέλει ήταν καλή η λύση. διότι φαίνεται ότι βοήθησε η εξέλιξη όλη αυτή τη γραμμή και βοήθησε την εξέλιξη όλη αυτή τη γραμμή. Δεν, δεν είμαι τόσο αρνητικό δηλαδή όσο στην αρχική μου τοποθέτηση. Για το δυναμικό υπάρχουν συζητήσεις για μια διπλή ε, ικανότητα δυναμικού. Ναι, το ξέρω. Αλλά εγώ θα αναφέρομαι σε μια μελέτη του Ινστιτούτου Επιστημονικών Μελετών της Τουτχάρδης που αναφέρεται σε μια αύξηση του δυναμικού κατά 30%. Δηλαδή, ο υπολογισμός είναι και ζήτημα μεθοδολογίας. Πώς αξιολογείται αυτή η ικανότητα, τι είδους ε, όγκο, τι είδους βάρος μπορεί να σηκώσει και εμένα με ενδιαφέρει φυσικά και περαιτέρω, ακόμα και αν δεν παραμείνω εγώ υπεύθυνο ε, στο έργο αυτό, θα το παρακολουθήσω. Βέντλιγκερ Ούλμ, ναι, όντως, χωρίς μεταφορά εμπορευμάτων, δεν αξιοποιείται η γραμμή τόσο όσο εάν είχαμε και τη μεταφορά εμπορευμάτων. Και το μόνο που μπορώ να κάνω να εκφράσω την ελπίδα αυτή η γραμμή Εάν μετατραπεί σε μια πολυτροπική γραμμή, Ρήνου, Δούναβη και το καθεξής, να ασχοληθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναπτύξει τη διάσταση της μεταφοράς των εμπορευμάτων. Βγαίνει. Εγώ με θαυμασμό σημειώνω τις καλές εξέλιξεις στο σταθμό. Τα δύο Άλλα γειτονικά κράτη δεν έχουν λάβει πέραν της Σλοβακίας οριστική απόφαση για τη γραμμή. Υπήρχαν κάποιες εναλλακτικέ, αρχικά τουλάχιστον είχαν προταθεί αρκετέ. Θα επιλεγεί κατά πάσα πιθανότητα η πιο βόρεια γραμμή. Αλλά, όπως είπα, αναμένεται και μια στρατηγική μελέτη από πλευράς Σλοβακίας. Όπως είπα, έχω συνομιλήσει με τον αρμόδιο υπουργό και αναλόγως αποφασίζουμε εάν το τούνελ αν η σύραγγα κάτω από το Δούναβι δηλαδή θα αποφασιστεί τελικά να κατασκευαστεί, εάν θα προτιμηθεί η λύση του αυτοκινητοδρόμου και μια, μια γρήγορη γραμμή συγγνώμη σιδηροδρομική ώστε να ε, συνδεθεί η ε, Βιέννη με την Πρατισλάβα και αντίστοιχα να ε, επεκταθεί και το αεροδρόμιο της Πρατισλάβα μετά. Μέχρι το 2020 τι θα έχει ολοκληρωθεί και τι όχι. Εγώ από το 2005 κρατάω στα πρακτικά μου ένα πολύ σημαντικό έγγραφο με υπογραφές τεσσάρων υπουργών μεταφορών που όριζαν ως στόχο για ολοκληρώση το 2016, ώστε να είναι ολοκληρωμένη ολόκληρη η γραμμή, μακροπρόθεσμα, έργα κτλ. Ε, μπορεί κανείς να ονειρεύεται, έστω και αν δεν μπορεί να τα υλοποιήσει όλα. Τώρα, μια ολόκληρη σειρά, γιατί έχουμε 22 τμήματα, σε 22 τμήματα χωρίς τη γραμμή αυτή, και για το κάθε ένα από τα τμήματα έχω νέες χρονολογίες, νέους στόχους. Το 20 λοιπόν. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο τουλάχιστον τμήμα της γραμμής αυτής θα είναι στη λειτουργία για τα υπερσυνοριακά ε, κομμάτια. Ναι, μπορεί να προσφέρει βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράδειγμα, η γέφυρα στο Κέλ και με πρόσθετη ε, υποστήριξη και ενθάρρυνση από την Ευρώπη μπορούμε να ε, ενθαρρύνουμε δύο μεγάλα κράτη-μέλη, μπορέσαμε να ενθαρρύνουμε δύο μεγάλα κράτη-μέλη να κατασκευάσουν αυτή τη γέφυρα. Για την Πρατισλάβα, όπως είπα, δεν υπάρχουν ε, πολιτικά εμπόδια, ούτε καν χρηματοδοτικά λείπει η απόφαση για το τεχνικό κομμάτι μόνο. Και τώρα στα κλικά. Σας ευχαριστώ για, για τα ερωτήματά σας. Ε, τις συμβουλές πρέπει να δώσω στους επόμενους που θα αναλάβουν αυτό το έργο. Το έργο προτεραιότητας 17 θα ενσωματωθεί ε, στον πολυτροπικό ε, διάδρομο Στρασβούργου-Σούλιναρ και στην Μαύρη Θάλασσα. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση γιατί δεν θα έχουμε μόνο μία απευθείας γραμμή, αλλά ένα σύνολο γραμμών και δύο παλιά κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν, Γερμανία-Αυστρία, αλλά και την πλειονότητα των σχετικά νέων ε, κρατών μελών. Εντάξει, βεβαίω έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία για το καθεξής. Επομένως έχουμε και τις παλιές αγορές και τις νέες από, τις, ε, από τα νέα κράτη-μέλη. Ο νέος ε, συντονιστής κατά πόσο θα μπορέσει να εκπροσωπήσει τη χώρα του. Εγώ θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου ε, σε άλλους τομεί, όμως τρία είναι τα κύρια μηνύματα τα οποία θέλω να αφήσω βάσει της ε, εμπειρίας μου. Πρώτον, εξέταση των εναλλακτικών προτάσεων. με κάθε σεβασμό προ την ε, αρχή τη επικορικότητας και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, μεγάλη εντύπωση μου είχε κάνει η πρώτη επίσκεψή μου στη Στουτγάρδη το 2005. Και πραγματικά θεώρησα εξαιρετικά εντυπωσιακό αυτό το σχέδιο ε, να αλλάξουν πολλά πράγματα για αυτό το σιδηροδρομικό σταθμό. Εγώ εξέφρασα ένα ιδιαίτερα τεχνικό ερώτημα προ του Γερμανού ομολόγου μου. ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσει που έχετε εξετάσει. Έλαβα την απάντηση, κανένα Alternative, καμία εναλλακτική. Ε, την αποδέχτηκα αυτή την απάντηση, όμως στην πολιτική όπως και στα τεχνικά ζητήματα πάντα υπάρχει και άλλη λύση, τουλάχιστον μία, αν όχι πολλές. Ναι, ποτέ δεν το επέκρυψα αυτό. Το επαναλαμβάνω τώρα μπροστά σε αυτό το πολυπληθές και ενδιαφέρον κοινό. Επομένω, το πρώτο μου μήνυμα είναι οι εναλλακτικέ λύσεις. Πάντα. Μετά, ε, εκτίμηση κόστους. Εδώ μπορώ να αναφερθώ σε πολλά τμήματα και να μην αποκλείσουμε εδώ και το Στουτγάρδι 22, γιατί σε αυτούς τους τομείς ποτέ δεν έχουν μειωθεί οι δαπάνες. Πάντα αυξάνονται. Το δεύτερο είναι αυτό. Και τρίτον, υπάρχει ένα μαγικό σημείο όπου μπορεί να αλλάξει η δημόσια στήριξη. Πότε δεν ξέρουμε πότε και γιατί, αλλά αυτό συνέβη και με τη Στουτγάρδη. Πέρα από τα πέντε δις, μετά είπαν όχι. Δεν δεχόμαστε αυτή την τιμή. Και μετά συνεχής αξιολόγηση κινδύνου συμπεριλαμβανομένη και της ε, δημόσιας στήριξη. Ποτέ να μην φυσικάζουμε. Ε, Με ένα project βέβαια κάθε χρόνο να επαναλαμβάνεται κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα μάθημα για όλους τους ε, πολυτροπικούς διαδρόμους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλάτς, για το έργο σας και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σέτσι. Mr. of course, is the... Ο κύριος Σέτσι είναι συντονιστής των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών για το έργο προτεραιότητας 3 και 9 που συμπεριλαμβάνει ένα από τα αγαπημένα μας προγράμματα το Figure Rest Α, το 9 εννοούσα. 3 και 19 μάλλον. Τα Γαφινιόν Φιγκέρες. Τα αγαπημένα μας έργα, έχετε το λόγο. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που περιβρίσκομαι εδώ σε αυτήν την Επιτροπή για αυτό το ραντεβού, το έγκυρο που έχουμε, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο, όταν προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση, να εντοπίζουμε τα ανοιχτά ζητήματα και ίσως να βρούμε και νέες βάσεις πρόοδου. Βέβαια αυτή είναι και μία ειδική συγκυρία, γιατί βρισκόμαστε στο τέλος ε, της ε, τρέχουσας προσέγγισης ε, ως προς τον προσδιορισμό έργων προτεραιότητας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και είμαστε στην αρχή μιας νέας προσέγγισης βάσει των διαδρόμων της, του νέου μέσου σύνδεσης της Ευρώπης Connecting Europe Facility που εγκρίνατε πριν λίγες ημέρες και σας ευχαριστούμε φυσικά όλους για τις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει στο να προσπαθείτε συνεχώς να βελτιώνετε το πλαίσιο που έχουμε ενώπιον μας για τα επόμενα έτη. Σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη παρουσίαση χρησιμοποιώντας ε, δύο διαφάνειες σε σχέση με το που βρισκόμαστε και ποια είναι τα πιο επίγοντα προβλήματα και βεβαίως στη συνέχεια ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις ή να ακούσω τα σχόλιά σας. Μιλάμε εδώ για το έργο προτεραιότητας υπαριθμών 3 και το βλέπετε βασικά με κόκκινο χρώμα στη διαφάνεια και αποτελεί το σύνδεσμο ξεκινώντας από την Πορτογαλία και φτάνει στη Γαλλία μέσω της Ισπανίας και το έργο προτεραιότητας 19 που είναι η διαλειτουργικότητα στην Ιβρική Χερσόνησο. Και φυσικά αυτό συνδέεται στενά με το προηγούμενο και εδώ βλέπετε στη μέση των Πυρηναίων δύο βέλη που είναι το έργο προτεραιότητας 16 το οποίο όχι μόνο αφορά την κεντρική διέλευση των Πυρηναίων, αλλά και τη σύνδεση με την Νότια Ισπανία, με το Κάσερες. Και εγώ έπρεπε να προσδώσω προσοχή για να το πω έτσι, και έπρεπε να προσπαθήσω να προετοιμάσω το έδεφος για μελλοντικέ εξελίξεις. Βλέπετε εδώ κάποια μπλε αστέρια σε αυτή τη διαφάνεια και εκεί βλέπετε τις ε, πλέον προσφατές πρόοδους. Και πάνω αριστερά έχουμε το σύνδεσμο Tour Bordeaux, τον κόμβο του Bordeaux και κατόπιν ε, έχουμε και τη σύνδεση με τη χώρα των Βάσκων. Εγώ πρόσφατα επισκέφτηκα αυτά τα μέρη και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Βέβαια υπάρχουν και κάποια προβλήματα που συνεχίζουν να είναι εκρεμή, όμως είμαστε κοντά στη λύση. Έχουμε τώρα το σκέλος στην Ιβερική που προδεύει σε πλατφόρμα στην Εξτρεμαδούρα και στην Καστήλια και βλέπετε εκεί να υπάρχει ένας σύνδεσμος που λείπει. Θα το σχολιάσω σε λίγο και κατόπιν από την πλευρά της Μεσογείου, δεξιά. Έχουμε άλλη μια ικανοποιητική κατάσταση σε σχέση ε, με την παράκαμψη νήμου Πελιέ στη Γαλλία και κατέπινε το τμήμα ε, Βαλένσια όπου ε, σας ε, ανέφερα. Έχουμε το τμήμα που ενώνει το Φιγέρας με την Βαρκελόνη και ε, λειτουργεί εδώ, ε, εδώ για κάποια χρόνια αυτό το σκέλος και νομίζω πριν δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και η δική σας επιτροπή επισκέφθηκε αυτή την τοποθεσία. Και περιμένουμε ο σύνδεσμος αυτός να ολοκληρωθεί 100% και να είναι επιχειρησιακό. Ακόμα περιμένουμε την ευτυχή αυτή μέρα, οπότε θα είναι δυνατό το τρένο υψηλής ταχύτητα να φτάσει στη Βαρκελόνη και από την ε, Βαρκελόνη να συνεχίσει. Συνεχίζεται η δουλειά, αλλά βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσουμε. Λοιπόν, να σας αναφέρω τώρα τα τέσσερα κυρία σημεία όπου πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Καταρχήν, μια ερώτηση. Ποια είναι η πιο αποτελεσματική οδός για τα εμπορεύματα στο τμήμα του Ατλαντικού, στο σκέλος του Ατλαντικού, λαμβάνοντας και υπόψη ότι ένα από τα σημεία αφετηρίας πέρα από τα λιμάνια της ε, Πορτογαλίας είναι το Αλγασίρα στην Νότια Ισπανία. Και προκειμένου να, και μάλλον πρέπει να καταστήσουμε αποτελεσματικό αυτό το σύνδεσμο για αυτό το σκοπό. Τώρα και πάλι σε αυτή την περιοχή, κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε, έχει να κάνει με το σχεδιασμό για την ολοκλήρωση ενός ε, συνδέσμου που λείπει, Εύωρα Κάι. Πρόσφατα είχαμε διαπραγματεύσεις για την περίοδο 2014-2020 για την πολιτική συνοχής Εκεί είχαμε κάποια καλά ποινήματα. Νομίζω ότι έχει προσδιοριστεί μια λύση. Όμως δεν έχει σημειωθεί ακόμη πραγματική πρόοδος επιτόπου. Συνεπώς, βλέπετε εκεί το πρόβλημα με μπλε στο χάρτη. Να έχουμε ένα πραγματικό και αποτελεσματικό σύνδεσμο μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας και πρέπει να βρούμε μια λύση στα θέματα αυτά. Το αργότερο, μέσα σε δύο χρόνια μέχρι το 2015. Ένα άλλο σημείο ανησυχία ε, αφορά την ένταξη των λιμένων στο διάδρομο της Μεσογείου. Συνεχίζονται οι εργασίες ε, ε, κατά τη διάρκεια του, κατά τμήμα του διαδρόμου. Υπάρχει εκεί το θέμα της λειτουργικότητας. Ε, θα πρέπει να έχουμε την εφαρμογή του διαδρόμου στη Μεσόγειο, όμως και εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Και πάνω απ' όλα το πιο σχετικό ζήτημα, σκοπιά ζήτημα, είναι πώς να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη διαλειτουργικότητας ε, στο σκέλος της Μεσογείου, κυρίως σε ό,τι αφορά το τμήμα Μομπελιέ Περπινιάν, που το βλέπετε με πράσινο δίπλα στο ερωτηματικό διαλειτουργικότητα. Και αυτό εμποδίζει την πλήρη εκμετάλλευση τη σύραγα και όλη τη δουλειά που έχει γίνει από τη Βαρκελόνη μέχρι τα γαλλικά σύνορα. Τώρα, να στραφώ και σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τον εγγύς μέλλον. Εδώ έχουμε δύο διαδρόμους, το ένα τηλεδικό διάδρομο με κίτρινο και ένα τμήμα του διαδρόμου της Μεσογείου με πράσινο. Τα βλέπετε σε αυτό το χάρτη. Γνωρίζετε βέβαια τα χαρακτηριστικά, πολυτροπικότητα κτλ. Και στην πράξη, όπως είπα, το έργο προτεραιότητας 3 και το έργο προτεραιότητας 19 θα συμπεριληφθούν πλήρως στους δύο νέους διαδρόμους που θα έχουν και ένα τμήμα από κοινού το οποίο το βλέπετε στο χάρτη μεταξύ, μεταξύ Αλχεσίρας Μαδρίτης. Και μετά τη Μαδρίτη έχουμε στροφή είτε προς τον Ατλαντικό είτε προς την Μεσόγειο. Ο μεσογειακός διάδρομος θα είναι ο πιο σημαντικός ε, για τη σύνδεση της Νοτιάς Ευρώπης, ε, Δύσης Ανατολής ε, και θα έχουμε και ένα νότιο διάδρομο Έχουμε την ε, Βόρεια Μεσόγειο, τη Σκανδιναβική, συγγνώμη, την Ανατολική πλευρά ε, του διαδρόμου της Μεσογείου. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικός ο ρόλος για να συνδεθεί η Νότια Δυτική Ευρώπη με την Ανατολική Ευρώπη μέχρι την Ουκρανία, αλλά και έχουμε και σύνδεση Βορρά-Νότου και ο Ατλαντικός διάδρομος φτάνει από το Ολχεσίρας στη Λεάβρα, στη Χάβρη στην Γαλλία και το Benelux ε, είναι ο κύριος κόμβος και θα συμπληρωθεί εκεί το τελικό τμήμα του έργου προτεραιότητας 17 στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μπάλατς. Αυτό είναι το τμήμα μεταξύ Παρίσιου, Στρασβούργου και στη Γερμανία στη συνέχεια. Σημαντικές ε, συνιστώσεις του διαδρόμου, ναι, ναι, ολοκληρώνω. Θα είναι η θαλάσσια συνιστόσα, έχουμε και τους αυτοκινητρόδρομους της θάλασσας και διαδρόμους εσωτερικής ναυσιπλοείας, επομένως ε, θα έχουμε ένα διάδρομο πλήρη, έτσι όπως το γνωρίζετε. Νομίζω ότι μπορώ να ολοκληρώσω εδώ, Πρόεδρε γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολλά σχόλια και παρατηρήσεις. Και σας έχω δώσει όπως και να έχει και τη γραπτή έκθεση. Ευχαριστούμε, Σάντερ και κύριε Σβίτα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Σέκη για τη σαφηνιά του και για την προσοχή με την οποία προετοίμασε τα συμπεράσματα. Επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί έχει λάβει υπόψη και την ε, εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει τονίσει και το άνοιγμα του Κανφρέν και νομίζω ότι είναι δύο σημαντικά θέματα αυτά τα οποία δυστυχώς ε, δεν έχουμε χρόνο να τα γιατί εκεί έχουν καταρρεύσει αυτά τα τμήματα λόγω προβλημάτων επιβατική σύνδεση. Τώρα, για τον διάδρομο της Μεσογείου. Εσείς ε, αναφερθήκατε σε αυτό με σαφήνεια, όμως το πρόβλημα σύνδεσης μεταξύ ε, Μονπελιέ και Νίμε. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα ε, γιατί πώς ε, θα κλείσουμε τα προηγούμενα έργα ε, αν υπάρχουν προβλήματα με το χρονοδιάγραμμα. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα έχουμε ένα πρόβλημα όχι μόνο εφαρμογής, αλλά και ένα πρόβλημα σύγκρουσης μεταξύ σχεδιασμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, υπάρχουν πολλές ανησυχίες ε, για τη σύνδεση Βαρκελόνης-Βαλένσια και από τη Βαλένσια και κάτω για το ποια τμήματα θα μπορούν να διατηρηστούν. Προβλέπεται μια διπλή πλατφόρμα και ε, τρίτη συνδρομική γραμμή που είναι μια ενδιαφέρουσα λύση και μας έχει επιτρέψει να υπάρξει πίεση. Όμως ε, στο μέλλον πώς θα διαμορφωθεί αυτό, αν μπορείτε να μας το προσδιορίσετε για τον Ατλαντικό διάδρομο. Σας ευχαριστώ γιατί ήταν ε, καλή πρακτική που ακολουθήθηκε στο Tour Bordeaux Όμω στην περίπτωση τη Πορτο... της Πορτογαλίας θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Βλέπω ότι εσεί σε έναν ε, σύνδεσμο πουλίτη για τη σύνδεση με τη Λισαβόνα και αντίθετα ε, φαίνεται να προτείνει η Πορτογαλία να υπάρχει μια σύνδεση με τη Σαλαμάνκα. Την επόμενη συνάντηση των συντονιστών πιστεύετε ότι μπορούν να υπεργαστούν καλύτερα με τον κανονισμό που έχει υιοθετηθεί. Ευχαριστώ κύριο Ζρικέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο οποίο συνδέεται με τα όσα ανεφερεινές, ε, κάνατε κάποιες προβλέψεις για τη σύνδεση Περπινιό-Μομπελιέ που δημιουργεί πρόβλημα. Ιδίως ότι φορά αυτό το ζήτημα με την νήμα. Και δεύτερον, έχετε αντίστοιχε προβλέψεις για τον Μπογντό Μπαγιόν και χώρα των Βάσκων. Είχατε δυνατότητα να το συζητήσετε, έχετε εσείς κάποιες ε, προτάσεις ε, ε, ότι πρέπει να γίνει μια επιλογή Μπορντό-Τουλούς και όχι Μπορντό-Ισπανία. Και οι απόψει ε, δίστατο ό,τι αφορά τα εθνικά συμφέροντα και βεβαίως ε, την ευρωπαϊκή διάσταση. Ποια είναι η σύνδεση λοιπόν μεταξύ αυτού του συνδέσμου που λείπει. Ευχαριστώ. Κύριε Μπιλμπάου, ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Σακή για τις εξηγήσει και κυρίως για την έκθεση που μας έχει στείλει. Θα επικεντρωθώ σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και μάλιστα αναφέρεται και στην έκθεση του κυρίου Σέκη για το Ατλαντικό διάδρομο. Στην έκθεσή σας τονίζεται ένα πρόβλημα που εμείς ως, πολιτική, ως πολιτικό κόμμα το έχουμε καταγγείλει σε διάφορους θεσμούς στο Ισπανικό κράτος αλλά και στις σχέσεις που έχουμε με τους Γάλλους ηθήνοντες. Όμως εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που είναι ο κόμβος της Μπεργκάρα που επιτρέπει να εφαρμοστεί όλα όσα έχουν εκτελεστεί αυτή τη στιγμή στο τμήμα του Ατλαντικού Διαδρόμου και κυρίως ό,τι αφορά στη χώρα των Βάσκων που θα επιτρέψει τη σύνδεση με τη Γαλλία. Εσείς έχετε συζητήσει με τους διάφορους συθήνοντες και ποια λύση πιστεύετε ότι θα πρέπει να βρεθεί τους επόμενους μήνες ή έτη, γιατί από την πλευρά της Ισπανικής Κυβέρνησης και του Ερμοδίου δεν υπάρχει καμία απάντηση ούτε για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτού του έργου, και βάσει των αντικειμενικών δεδομένων ε, και των ε, προπολογισμών που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει σοβαρή δέσμευση από την Ισπανική κυβέρνηση για να εκτελέσει αυτό το τμήμα του έργου. Επίση, εδώ βλέπουμε ακριβώ με κόκκινο τα δύο τμήματα των συνόρων και να σα ρωτήσω λοιπόν με αυτή την έκθεση που εκπονήθηκε ε, από διάφορους Γάλλους ε, ηθήνοντες όπου δεν τέθηκε με καθοριστικό τρόπο η υλοποίηση κάποιων ε, έργων προτεραιότητα που εγκρίναμε στην Λομέλεια. Πώς εξελογείτε εσείς την κατάσταση και τι μπορούμε να κάνουμε για να πείσουμε τα κράτη ότι τα ευρώ που έχουν στον προπολογισμό πρέπει να κατευθυνθούν προς τα έργα προτεραιότητας αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει σύνδεση και αν θέλουμε να θέσουμε τέλος σε αυτά τα σύνορα που συνεχίζουμε να έχουμε και θα, μάλλον θα συνεχίσουμε να έχουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα από μένα. Κατόπιν τα όσα είπαν και Ρίκια και Βιλμπάου. Υπάρχει εδώ ένα θέμα, μια σύγκρουση μεταξύ εθνικών συμφερόντων ιδίως των γαλλικών, σε ό,τι αφορά τους διαδρόμους. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το πρόβλημα. Για μένα είναι εξαιρετικό που μπορούμε να, να πάμε από το Φιγκούρα σε, στην Περπινιόν. Είναι εξαιρετικό. Όμως δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Εάν δεν υπάρξει η συνδεση ή Μομπελιέ-Περπινιόν. Βεβαίω, εντάξει, εγώ δεν είμαι αντικειμενικό, γιατί λατρεύω το Περπινιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την τελευταία. Έχουν διατυπώσει και άλλοι βουλευτές. Ξεκινώ με δύο λόγια πρώτα. Δύο μόνο, αλλά σημαντικά. Συμφωνώ με την κυρία Πιλπά ότι πρέπει να αξιοποιούνται τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά, στο μέγιστο δυνατό βαθμό να υπάρχουν κίνητρα για να κατευθύνονται οι αποφάσεις. Και όλα αυτά βεβαίως πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό συμφέρον και την προσθέμενη αξία. Πρέπει ακόμα να προσπαθήσουμε για βελτίωση και βελτίωση και βελτίωση. Για το Περπινιά Φιγκέρας. Διασύνδεση κύριο πρόβλημα είναι η διαλειτουργικότητα στη Γαλλία. Στο κομμάτι του Πενιάκου Μομπελιέ, όπου εντοπίζονται προβλήματα που θα χρειαστούν χρόνο για να λυθούν και από ταυτόχρονα μπορούν να δουν και μεταβατικές λύσεις. Ξέρω ότι και από την ισπανική και από τη γαλλική πλευρά γίνονται οι σχετικές προσπάθειες. Και έρχομαι σε δύσκολη θέση, αλλά θα σας πω ότι δεν μπορώ να έχω μια σαφή εικόνα του πότε επιτέλους θα εγγενιαστεί η υπηρεσία αυτή η σιδηροδρομική χωρίς να χρειάζεται μεταπιβίβαση. Και βρίσκομαι σε μηχανή όπως είπα, γιατί, γιατί έχουν γίνει ανακοινώσει οι οποίες έχουν ανακληθεί, έχουν αναιρεθεί. Τελευταία, από την Ιταλική, από το Ιταλικό Σιδηροδρομικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Ιταλικό Σιδηροδρομικό Πρακτορείο Ειδήσεων και αναφερόταν στις 15 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή. Οι Ισπανοί όμως θα τους ρωτήσουν να μας είπαν να δεν έχουμε ιδέα. Άρα ναι, έχετε δίκιο. Κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να ασκηθεί ακόμη περισσότερη πίεση για τέτοιου είδους καταστάσεις. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει και υπόδειγμα για το μέλλον. Γιατί είναι δύσκολο να δεχθεί κανείς τόσα χρήματα να ειστρέουν σε τέτοιου είδους έργα με έμπλοκη και ιδιωτών, ε, επενδυτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, εάν δεν προχωρήσει όλη η υλοποίηση με βάση το σχέδιο. Καθώς δε και λόγω της σπάνιδας κονδυλίων προσπαθούμε ιδιαίτερα να ενισχύσουμε τη διάσταση των ΣΔΙΤ, συμπράξεων δημοσιογραφικού τομέα, όποτε υλοποιείται ένα ενδιαφέρον τέτοιο έργο. Προσπαθούμε να προωθήσουμε την θέση σε λειτουργία του κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Για φανταστείτε δηλαδή το πιο σπουδαίο από αυτά τα έργα. Τουρ Μπορντό. Για οποιοδήποτε λόγο να αντιμετώπισε προβλήματα και δεν θέλω να φανταστώ τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ασκήσουμε τις πιέσεις στους εμπλεκόμενους φορείς, στους και κυβερνήσεις. Και έτσι προχωρώ και στα λοιπά ερωτήματα. Η κεντρική διάβαση που είναι περιλαμβάνοντας στο συλλογικό δίκτυο. Και αυτό γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2030, ίσως το 2050. Και πάντως δεν, παρά, δεν θα ήταν ούτως ή άλλως ε, επιλέξιμο, παρά μόνο για μελέτες, σχεδιασμό κτλ. Και μετά θα έπρεπε να διατεθούν κονδύλια και ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση πιο αποτελεσματική και ταχεία για την υλοποίηση του. Χρονική ορίζοντας δεν είναι κάτι άλλο. Άλλο έργο θα τελειώσει στα 10 χρόνια, άλλο στα 20, άλλο θα το δουν τα εγγόνια μας. Τούτου λεχθέντος Ας ρίξουμε μια ματιά και στην άλλη πλευρά τον Ατλαντικό και την ερώτηση της κυρίας Μπιλμπάου. για το πώς αντιλαμβάνομαι, τι γνώμη έχω για τη στάση της γαλλικής κυβέρνησης. Ξέρετε ότι η Κομισιόν Μομπιλιτέ 21, η Επιτροπή για την Κινητικότητα, ε, κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα προ προς το γενικό σχεδιασμό έργων υψηλής ταχύτητας που θα πρέπει να υλοποιηθούν στη Γαλλία. Θα ξέρετε ασφαλώς όμως και ότι ο υπουργό Κουβιέ είπε πως η διασύνδεση με την Ισπανία, Μπορντό, Ενάι και Τουλούζη που εξασφαλίζει τη μετάβαση από τον Ατλαντικό στη Μεσόγειο ακόμη είναι στο στόχαστρο της γαλλικής κυβέρνησης. Ακόμη είναι στόχος της γαλλικής κυβέρνησης να ολοκληρώσει αυτό το έργο, έστω με κάποια επιβράδυνση λόγω των δυσκολιών, γιατί τώρα προσπαθούν να βελτιώσουν την υφιστάμενη γραμμή Μπορντό Εντάια, που έχει πολύ περιθώριο για βελτίωση. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοινώνει ότι σε δύο-τρία χρόνια ή και το 2018 θα είναι σε πλήρη λειτουργία το ΙΕΝΤ για το γαλλικό στο δρομικό δίκτυο, στο σύνολό του, κάτι το οποίο βρίσκω πολύ, πολύ σημαντικό, ακόμα και νωρίτερα μπορεί να συμβεί. Και έτσι έχουμε μια βελτίωση, έστω και σε προσωρινή βάση, μέχρι να γίνει η καινούρια γραμμή. Πάντως η διασύνδεση στα δίκτυα υπάρχει. Στην πρόσφατη μου επίσκεψη είδα μια σαφή ένδειξη ότι έχει γίνει αντιληπτό το πρόβλημα και ότι θα δοθεί λύση. Ιδιαίτερα λαμβανωμένο η υπάγωψη του γεγονότο ότι από τώρα έως το 2018 θα έχει ολοκληρωθεί το βασικό δίκτυο για να φτάσει μέχρι τα σύνορα και με ένα ενδιαφέρον σχέδιο για την παράκαμψη του Σαν Σεμπαστιάν. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Από τη Γαλλία έως το 2018 και έτσι μπορούμε ίσως να έχουμε πλήρη εκμετάλλευση του νέου δικτύου από εκεί και πέρα. Η δε συμφόρηση που υφίσταται, γιατί τη συμφόρηση βέβαια την έχουμε τώρα σε οδικές μεταφορές, και αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη του πόσο επίγον είναι να προχωρήσουμε σε μια αναλλακτική η οποία θα προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων σιδηροδρομικός και επίσης θα έρθει η ώρα να δούμε και εκεί τη συμφόρηση και το θέμα των κεντρικών διαβάσεων. Νομίζω ότι τα έχω καλύψει όλα. όσα με ρωτήσατε. Δύο-τρία λόγια μόνο για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Για την δέσμευση. Για τη διακυβέρνηση και το PP3. Πορτογαλία, Ισπανία. Η ε, Γαλλία. Είδαμε πριν από μερικέ ημέρε και ήσασταν νομίζω κάποιοι παρόντε την ε, υπογραφή για μια δέσμευση για τον Ατλαντικό διάδρομο από τους τρεις υπουργούς ή υφυπουργούς αναλόγως που ήταν εκεί παρόντες. Ένα έγγραφο που δεν περιορίζεται σε μια δήλωση στον τύπο, αλλά δεσμεύει κυβερνήσεις. Και μια τελευταία παρατήρηση. Υπάρχουν ασφαλώς οικονομικά προβλήματα. Όταν ανοίξει νέα φάση θα συνεχίσουμε παράλληλα με αυτήν να επαγρυπνούμε για να αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο τις οικονομικές διαστάσεις. Για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη χρήση των PPP, τη χρήση των ομολόγων έργου, Και θα συνεχίσουν βέβαια και οι ιδιωτικοί ε, πάροχοι στις διάφορες χώρες, Ισπανία, Ιταλία κτλ. την εξέταση των βέλτιστων δυνατών πρακτικών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σέκη. Ο κύριος θα έχει αργήσει. Άρα παρακαλώ τον κύριο Βίνκ. Κάρελ. So, ERTMS, Carol, floor is, is yours. I'm just about on time. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω και εγώ να τηρήσω το χρονικό όριο. Σε ό,τι αφορά το EMS, θεωρώ ότι είμαστε πιο αισιόδοξοι φέτος σχέση με πέρυσι. Έχουμε δύο πρότυπα, το 230 Δέλτα, το οποίο ήταν έτοιμο το 2008 και το άλλο και το κυριότερο, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2012. Άλλη σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά το σύστημα διαχείρισης ε, είναι η γενικότερη ατμόσφαιρα και η απόφαση της Γερμανίας. Και πλέον είμαστε πεπισμένοι ότι είναι το ένα και μοναδικό σύστημα σηματοδότησης στην Ευρώπη. Έχω πει πολλέ φορέ ότι φορά τη διαλειτουργικότητα και οι άλλοι συντονιστέ ανέφεραν ότι σε ό,τι αφορά τη διατροπικότητα υπάρχουν τρει όροι που πρέπει να πληρούνται. Ένα, ότι πρέπει να αφαιρεθούν ε, τα σημεία ε, συμφόρησης από τις υποδομές, μετά ε, η εισαγωγή του ΙΑΤΜΕΣ, e του προτύπου και η αναρμόνιση των εθνικών κανόνων ασφαλείας. Τι συμβαίνει σήμερα. Και θα επιμείνω στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος που ανέφερε ο Πρόεδρος. Να σας δώσω κάποια κύρια σημεία για τις ε, δραστηριότητες μας στο μέλλον. Θέλω να επιμείνω ότι ίσως είναι καλύτερα να ξεχάσουμε το ERTMS ως όρο και να μιλήσουμε περισσότερο επί της ουσίας στην Επιτροπή μας. Σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα. Πρέπει να καταστεί διαλειτουργικό το σύστημά μας. Και σε ό,τι αφορά το πρότυπο, αποδεχόμαστε ένα ελάχιστο τροποποιήσεων γιατί έτσι περιπλέκεται το σύστημα, καθίσταται λιγότερο ασφαλές και είναι και πιο δύσκολος ο έλεγχός του. Πώς ακριβώς το κάνουμε αυτό. Θα εξετάσουμε συγκεκριμένα τα διασυνοριακά τμήματα, γιατί θεωρούμε ότι αν εξετάσουμε τα διασυνοριακά τμήματα ένα προς ένα ως έργα, ως project, αν δούμε 20, ακόμα και 10 εγώ θεωρώ τέτοια τμήματα διασυνοριακά που μπορούμε να εξετάσουμε και να λύσουμε ζητήματα μεταξύ παρόχων, ε, δικτύου και το καθεξής, τότε λύνουμε, 80 αν όχι 90% των προβλημάτων διαλειτουργικότητας. Θα δούμε λοιπόν τα διασυνοριακά τμήματα συγκεκριμένα και κατά τη γνώμη μου έτσι θα λύσουμε, όπως είπα, 80% των προβλημάτων διαλειτουργικότητας. Δεύτερον, ενίσχυση της υλοποίησης του ERTMS. Είχαμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ε, Deployment. Κάποια κράτη-μέλη παρουσιάζουν καθυστερήσεις και θα δούμε τι είδους μέτρα ή κίνητρα μπορούν να δοθούν για να επιταχυνθεί η εφαρμογή του συστήματος. Μετά, σε ό,τι αφορά την τυποποίηση, που ήταν και ένα από τα ζητήματα που με απασχόλησε περισσότερο, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση στην βασική γραμμή 3, baseline 3. Μόλις οριστικοποιηθεί από τον ΕΡΑ, θα δώσουμε αυτή τη βασική γραμμή στους τοπικούς μας φορείς. Τέταρτον, θα ήθελα να καλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο ρόλο του ΕΡΑ ε, στο πλαίσιο του τέταρτου πακέτου για τους σιδηροδρόμους. Είναι πολύ σημαντικό για την ε, γενικότερη εφαρμογή του προγράμματος λειτουργικότητας. Πέμπτον, υπάρχει και ένα θέμα με το σύστημα κοινοποίησης. Ξέρετε ότι είναι ε, τμήμα του ETCS, του συστήματος σηματοδότησης. Ξέρουμε ότι το υφιστάμενο σύστημα μπορεί να καταστεί παροχημένο μέχρι το 2022-2025. Θα δούμε λοιπόν τι θα αντικαταστήσει αυτό το σύστημα κοινοποίηση. Μία αρχή θα ακολουθήσουμε, σαφής διάκριση των συστημάτων. Το ETCS που έχει αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή ως Baseline 3 θα πρέπει να ε, επικοινωνεί με οποιοδήποτε άλλο σύστημα κοινοποίησης ενδεχομένως υιοθετήσουμε. Μετά, αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε αναπτύξει τώρα αναγνωρίζεται όλα και περισσότερο σε παγκόσμια κλίμακα ως ε, το κατεξοχήν ε, σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου ταχύτητας. Πρέπει να πιέσουμε αλλά και να στηρίξουμε την, τον κλάδο της βιομηχανίας ότι αυτό θα είναι το σύστημα το οποίο θα γίνεται αποδεκτό και θα εφαρμόζεται και από τεχνική ε, σκοπιά και σε ό,τι αφορά τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αυτά είναι τα κύρια σημεία, Πρόεδρε. Αν τα υιοθετήσουμε, έχουμε πρόγραμμα για τα επόμενα έτη και έτσι θα συμβάλλουμε τα μέγιστα σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητα, που είναι το πιο σημαντικό για μένα. Αν θέλετε να κρατήσετε ένα πράγμα από την ομιλία μου σήμερα, είναι το ζήτημα της διαλειτουργικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βίν και κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Βίνκ για την παρουσίασή του και για την ειλικρινιά του, γιατί μας είπε που βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα. Ε, τώρα, όπως ξέρετε, τώρα εμείς εργαζόμαστε εις βάθος το θέμα της λειτουργικότητας στο τέταρτο συνδρομικό πακέτο και έχουμε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα τα οποία ουσιαστικά σας αποδίδουν δίκαιο σε σχέση με τα προβλήματα που έχει ένα συγκεκριμένο κάτω μέλο. Θέλω να σας ρωτήσω εσείς τι συστήνετε να εξοπλιστούν ε, ε, τα τρένα μέχρι να περιμένουμε την προσαρμογή της υποδομής. Δηλαδή εσείς συστήνετε οι μηχανές των τρένων να αποκτήσουν αυτό το σύστημα ETCS και πόσο παραπάνω κοστίζει αυτό και αν αυτό ε, ε, σημαίνει ότι τελικά δεν είναι καλό το μήνυμα που δίνεται και θα εγκαταλείψουμε το σύστημα ERTMS. Η κυρία Μπιλμπάο, ευχαριστώ πολύ για όλες τις εξηγήσεις. Εργαζόμαστε εντατικά και θα δούμε τι θα συμβεί με όλη τη δεσμή μέτρων. Όμως ε, και εμείς εργαζόμαστε επί της έκθεσης για τη λειτουργικότητα και προσπαθούμε να συμβεστούμε τις προθεσμίες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη σε σχέση με το ρόλο του ΕΡΑ και τη σχέση με τους εθνικούς οργανισμούς. Εσείς θεωρείτε ότι ε, αυτή θα έπρεπε να είναι η αρμόδια για να αναλάβει όλα αυτά τα ζητήματα ή πιστεύετε ότι θα χρειαζόταν μια μεταβατική περίοδος και ποιο ρόλο θεωρείτε ότι θα έπρεπε να διαδραματίσουν ε, οι εθνικοί οργανισμοί προκειμένου να υλοποιηθεί η εφαρμογή αυτού του συστήματος και αν τελικά την απόφαση αυτή την υποστηρίζουμε και την έχουμε όντω λάβει, πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα που δεν έχουμε κάνει ακόμα. Ευχαριστώ κυρία Μάσινερ. Μια πολύ στομή ερώτηση και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. σας. Με πολύ χαρά σημειώνω ότι το RTMS δεν είναι πλέον πρόβλημα για τη Γερμανία. Είναι ένα ETMS light όμως, αν μπορώ να το πω έτσι. Αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Και υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα στις, σε άλλες χώρες και περιοχές. Κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λέω Ρικέ. Θα ήθελα στα πίσω του χρόνου που έχει ο κύριο Βίνκ να μας πει κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με τις δυσκολίες που υπάρχουν για την εξέλιξη μεταξύ του ETCS και του συστήματος επικοινωνίας. Είπε πως ε, θα έπρεπε να απαλλαχθούμε από τέτοια ζητήματα, αν μπορείτε να μπείτε σε κάποιε περαιτέρω λεπτομέρειε για το τι πρέπει να συμβεί στο μέλλον. Ο πρόεδρο. Ε, ευχαριστώ. Να πω κι εγώ δύο λόγια. Θυμάμαι να πω τη σκοτεινή εποχή που προσπαθούσαμε να κάνουμε τα κράτη-μέλη να δεκτούν το σύστημα διαχείριση τη κυκλοφορία ε, και άκουσα ότι και η κυρία Μάισνερ ότι τώρα ε, η Γερμανία ε, βλέπει το πράσινο φως ότι αφορά το RTMS, όμως υπάρχουν χώρες όπου δυσκολευόμαστε και στο Ηνωμένο Βασίλειο δυσκολευόμαστε να σημειώσουμε πρόοδο. Ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με το RTMS στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεύτερον θέλω να σχολιάσω και το θέμα του συνδρομικού πακέτου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η τεχνική πυλώνες του τέταρτου πακέτου και κάποιοι, όπως και εγώ, πιστεύουμε ότι είναι το πιο σημαντικό τμήμα το ε, θέμα της διαλειτουργικότητας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο Κάρλ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις διάφορες ερωτήσεις ε, που έχουν τεθεί. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό των ε, μηχανών. Εγώ θα περίμενα ότι μέσω της τυποποίησης του baseline 3 επί του τρένου θα έχουμε πιο αποτελεσματικό σύστημα και λιγότερο δαπανηρό. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα, ιδίω στην Ισπανία, γιατί έχετε το baseline 2. επί πρέπει, αν τελικά καταλήξουμε σε αυτήν την απόφαση ότι το baseline 3 θα είναι εξοπλισμό που θα πρέπει να έχουν ε, τα τρένα, οι μηχανές, τότε θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η μετάβαση από το σημερινό σύστημα με το baseline 3. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα ήταν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αν μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό επί του τρένου στο baseline 3 γιατί είναι πραγματικά ευέλικτο το σύστημα και έχει συμβατότητα ε, και με την δομή baseline 2 που υπάρχει στην Ισπανία και με την ε, υποδομή baseline 3. Επομένως αυτό δεν έχει καθοριστεί ακόμα, αλλά έχουμε κάποιες ιδέες ε, για το αν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο και το έχω συζητήσει και με τη βιομηχανία και αν καταστεί δυνατό τότε θα τους ωφελήσει όλους και τους σιδηροδρόμου και φυσικά τη βιομηχανία τώρα σε σχέση με το ρόλο των εθνικών οργανισμών και τον αέρα. σε σχέση με τα όσα υπάρχουν στο τέταρτο συνδρομικό πακέτο και με το οποίο πρέπει να συμφωνήσετε, νομίζω ότι εκεί οι αρχές είναι καλές. Όμως το πρόβλημα είναι το εξή. Πρέπει να δούμε ποιο είναι ο ρόλο των NSA σε σχέση με το ρόλο του ΕΡΑ. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο ΕΡΑ θα είναι αρμόδιος ε, για όλες ε, τις διαδικασίες έγκρισης ε, σε κάθε χώρα. Θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των εθνικών αρχών ασφαλείας και του ΕΡΑ. Όμως, στο τέταρτο πακέτο προτείνεται ότι η αρχή που θα είναι αρμόδια να καθορίσει το πώς θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα αυτά και που θα έχει την ευθύνη είναι η ΕΡΑ. Θα πρέπει να έχει κάποια εξουσία, κάποια αρμοδιότητα και πρέπει να προσδιορίσουμε ποια θα είναι αυτή. Έτσι λοιπόν ε, στις διαδικασίες έγκρισης θα περιορίσουμε το ρόλο των εθνικών οργανισμών και θα αυξήσουμε το ρόλο της ΕΡΑ. Τώρα το πού θα ευρεθεί η ισορροπία θα συζητηθεί τους επόμενους μήνες. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για τις άλλες χώρες, μπορώ να πω ότι με ικανοποίησε η απόφαση της Γερμανίας ε, και Όλες οι επαφές που είχαμε μέχρι τώρα είναι θετικές. Επίσης έχουν δεχτεί ότι η προτεραιότητα για τους διαδρόμους, κυρίως αυτούς που εξετάζουμε υπό το φως των ευρωπαϊκών διαδρόμων, είναι ο διάδρομος Ρενού Άλπεν ή από το Ρότερνταμ στη Γερμανία και επομένω έχουν δεκτεί οι Γερμανοί και αυτή την προτεραιότητα και πραγματικά δεν μπορώ να παρεπανεθώ για τη στάση της Γερμανίας. Το αντίθετο, υπάρχει βέβαια ένα μικρό πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω και έχει να κάνει ε, με την ε, Γαλλία. Δηλαδή μπορεί να επιταχύνουμε τη διαδικασία αν αποκτήσουμε μια πιο στενή σχέση με το Γαλλικό Υπουργείο. Έχουμε πρόβλημα όμως να πείσουμε τις γαλλικές αρχές να προχωρήσουν με το πρόγραμμα το οποίο είναι τμήμα του σχεδίου ανάπτυξης και αν σκεφτούμε τις προθεσμίες αυτό θα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που θα πρέπει να συζητηθεί με τις αρχές. Για το Ηνωμένο Βασίλειο μπορώ να πω ότι η σχέση εκεί είναι διαφανής και ανοιχτή. Βεβαίως, όπως πάντα, έχει τι απόψει του το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όπως και να έχει υπάρχει ένας διάλογος και δεν έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν ε, έχει εφαρμοστεί όμως καθόλου τερδί μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, αλλά πρέπει να ξεκινήσει κανείς με το πρώτο και οι προσπάθειες που γίνεται για την επέκταση της γραμμής υψηλής ταχύτητας οδηγούν και στην υιοθέτηση του e RTMS. Είμαι όμως αισιόδοξο για το πώς μπορούμε να το χειριστούμε το ζήτημα για το σύστημα επικοινωνίας στο περιφερειακό Ρικέ. Το πρόβλημα είναι το εξή. Σήμερα το RTMS είναι ο συνδυασμό του ETCS συν το GSMR. Και το GSMR είναι σύστημα επικοινωνία που έχει αναπτυχθεί για του σιδηροδρόμου. σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων που θα χρειαστεί στο μέλλον και που δεν συνδέεται μόνο με το σύστημα έτοιμες, αλλά μπορεί να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη διαβίβαση δεδομένων για να λάβουμε υπόψη την αποτελεσματικότητα που θέλουμε στους δρόμους σε σύγκριση με τις σχετικές μεταφορές, με τις οδικές μεταφορές. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι ευρύτερα και μεγαλύτερα ως προς τη χωρητικότητα για τη διαβίβαση των δεδομένων. Και εδώ πρέπει να αποφασίσουμε ποιο σύστημα επικοινωνίας θα χρησιμοποιήσουμε, τι είδους ο πιο εύκολος τρόπος, κατά την άποψή μου, θα ήταν να έχουμε μια συμφωνία, να χρησιμοποιήσουμε το 3G ή το 4G, ένα παγκόσμιο σύστημα επικοινωνιών. Βέβαια, μπορώ να σας πω, κύριε Ρικέ, ότι για το χρονοδιάγραμμα έχουμε κατά νου το εξής. Μέχρι το 2018 θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει, θα προτείνουμε τι είδους σύστημα επικοινωνίας θα χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να προετοιμάσουμε φυσικά και την μετάπτωση στο νέο σύστημα και μετά μέχρι το 2022-2023 θα είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε αυτό το νέο σύστημα επικοινωνίας. Όμως ε, όλα αυτά είναι υπό εξέλιξη. Thank you very much, Mr. Vink. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίνκ. Ακόμα μια κουβέντα. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστώ τον Πρόεδρο και την Επιτροπή για όλη την υποστήριξη που προσέφεραν στο έργο αυτό. Πολλές φορές ήταν σαν τον ατέρα του λοχνέ, Αλλά έχουμε μπει στο σωστό δρόμο. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει και θα είναι αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα και τουλάχιστον για το χρόνο που έχω συντονιστεί σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Και κανονικά θα πρέπει να έχουμε τον κύριο Μπριγχόρστ ο οποίος είναι καθοδόν. Ας κάνουμε τρία λεπτάκια διάλειμμα. Μέχρι τις πέντε φαντάζομαι να έχει έρθει, αλλιώς θα έχουμε βγει τελείως εκτός προγράμματος. Μερικά λεπτά διάλειμμα για τον κύριο Μπριγχόρστ. Okay, colleagues. Συνάδελφοι, σώσαμε τον κύριο Βίνκορστ από τις ε, υπηρεσίες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι συντονιστής για το έργο 6, Λιόν, Τεριέστη, Βατσοκόπα, Λουμπλιάννα, Βουδαπέστη, Ουκρανία. Έχετε το λόγο. 7 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη στους ε, πρώην συναδέλφους ε, που καθυστέρησα. Όμως, για να μπει κανείς σε αυτό το εκτήριο, ακόμα και αν για πολλά χρόνια είναι ευρωβουλευτής ή ήταν στο παρελθόν ευρωβουλευτής, είναι πραγματικά αδύνατον. Και η διαφάνεια την οποία θέλουμε η οποία θέλουμε να υπάρχει πρέπει να ισχύει και σε αυτό το τομέα. Πρόεδρε, τώρα επί του ζητήματος για το σχέδιο 6. Έχω κάποια καλά νέα, γιατί στους, στα δύο τμήματα, τεριέστη Τιουάτσα και Λιών Τουράν, υπάρχει, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για τη Λιόν Τωρίνο κατά τη γνώμη μου είναι πραγματικά το πιο σημαντικό μεμονωμένο έργο ε, σε όλο τον ε, διάδρομο της Μεσογείου γιατί αφορά και όλες τις υφιστάμενες ε, διασυνδέσεις και από την γαλλική και την ιταλική πλευρά. Βεβαίως σύντομα θα έχουμε και την πολωνική και ισπανική πλευρά. Το τελευταίο χρόνο στην Ιταλία τα έργα στο, ε, στη σύραγα Λαμαντελένα ξεκίνησαν. Έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για να ε, ολοκληρωθεί μέχρι τα 2016, στα μέσα του 2016 κατασταθένατο το έργο, με ένα χρονικό περιθώριο τριών ετών. Πραγματικά ήταν ε, πολύ σημαντική ε, εξέλιξη και αναγνωρίστηκε και από τους ε, ε, από τον πρόεδρο Λάντι και τον πρωθυπουργό Λέτα στη συνοδοκορυφή. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα έργα που προχωρούν με πολύ σημαντική πρόοδο και αναμένεται τα έργα αυτά να παραχωρηθούν στις αρχές του 2014. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρώμη. Έτσι, έχουμε φτάσει στο σημείο δίχως επιστροφή. Τα ανακοινωθέντα τύπου δεν μιλούν πλέον για έργο, για project, για σχέδια, μιλούν για εργοτάξιο, για ένα έργο το οποίο προχωράει. Με τα χαράς μπορώ να σας πω ότι από τη γαλλική πλευρά έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και στη Βουλή και στη Γερουσία και στην Ιταλία πριν τα τέλη του έτους θα γίνει η ψηφοφορία στη Γερουσία. Και κατά πιθανότητα από την πρώτη πρώτου θα έχουμε πλήρη έναρξη όλων των δραστηριοτήτων. Πολύ θετικά λοιπόν όλα αυτά για ένα έργο το οποίο έχει γνωρίσει πολλές καθυστερήσεις και πλέον η εφαρμογή του είναι το κύριο σημείο, όχι το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει όχι. Προ... Σύντομα, Πρόεδρε, γιατί καθυστέρησα κιόλα για την Ιταλία-Σλοβενία. Έχει σημειωθεί η πρόοδος. Πλέον υπάρχει μια κοινή Ιταλοσλοβενική δομή που θα καταστεί επιχειρησιακή τον Ιούνιο μέσω ε, ενός φορέα που έχει έδρα την Τεργέστη και έχει δύο διευθυντές, ε, μία από κάθε χώρα. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε το προκατακτικό σχέδιο, βεβαίως με μελέτη περιβαλλοντολικού αντικτύπου και εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές. Από το παρελθόν έχουμε διδαχθεί ότι είναι πολύ σημαντικό να εμπλέκουμε όσους ε, υφίσταται, υφίστανται τις ε, συνέπειες και γνωρίζω τα πράγματα από πρώτο χέρι. Συμπεραίνω λοιπόν Πρόεδρε ότι για τα δύο κύρια project Τριέσι Ντιβάτσα και Λιών ε, Τωρίνο τα πράγματα βαίνουν καλώς. Βεβαίως θα μπορούσαν να είχαν γίνει και πιο σύντομα αλλά εφόσον και η κοινή γνώμη είναι ακόμα και εχθρική απέναντι σε τέτοια προγράμματα, αλλά και εξαιτία των δημοσιονομικών περιορισμών είναι σχεδόν θαύμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Που ελήφθησαν και τόσο δύσκολες αποφάσεις αυτά τα δύσκολα χρόνια. Πιο πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής του Νοεμβρίου. Γενικά λοιπόν παραμένω αισιόδοξο. Οι νέε κατευθυντήρε γραμμέ μαζί με το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη έχουν υιοθετηθεί και χάρη ε, στο εξαιρετικό έργο του Κοινοβουλίου θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε και ελπίζω ο διάδοχός μου να επωφεληθεί από, τις, ε, από την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για Αλεσάντερ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πινχόρστη για την ενημέρωση και να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που τα εμπόδια που προκαλούσαν την καθυστέρηση έχουν κατά κάποιο τρόπο έρθει. Θέλω να ρωτήσω αν ε, οι Ιταλικές αρχές έχουν σεβαστεί τη δεσμευσή τους για τη χάρξη και τι ε, γίνεται με το γαλλικό σχέδιο υποδομών που δεν προβλέπει τις εθνικές συνεισφορές για τη σύραγα τουλάχιστον μέχρι το 2030. Δηλαδή, πόσο εσείς πιστεύετε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία σας μπορείτε να βελτιώσετε τα χρονοδιαγράμματα γιατί θα ήταν ε, κάπως γελίο να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή την λειτουργία τους, της ε, σύραγας ε, και να μην υπάρχουν οι συνδέσεις με άλλες τοπικές περιοχές. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Ευχαριστώ. Την ίδια ερώτηση είχα και εγώ. Γιατί αν το έργο ήδη κοστίζει πάνω από 10 δις, ε, τότε έχουμε 20 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κόστος ε, για ε, το έργο σύνδεση τη Λιών με τι υπόλοιπε τοποθεσίε. Και δηλαδή τελικά τι θα κάνουμε, θα κατασκευάσουμε μία σύραγα χωρί να την συνδέσουμε. Και τι θα γίνει με τη σύνδεση μεταξύ Λιών και Σύραγας. Δεν μιλώ καν για την παράκαμψη της Λιών που ήταν ένα συστατικό μέρος του σχεδίου. Και ε, βλέπουμε ότι έχουμε τελικά ένα έργο όπως είναι αυτό το οποίο το βάζουμε στη μέση του πουθενά. Ευχαριστώ κύριε Ρίκε. Και εγώ να πω δύο λόγια. Ανησυχώ κάπως για το σύνδεση της Ιταλίας με τη Σλοβενία και με τη σύνδεση με το λιμένο της Κόπα. Γιατί βλέπουμε ότι εδώ πρέπει να αρχίσουν οι εργασίες μεταξύ 2013 και 2015. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι έργα γίνονται συγκεκριμένα στη Σλοβενία, από τη σλοβενική πλευρά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να πατήσω στην κυρία Γιάλα Σέντερ. Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδρομή, υπάρχει πλήρη συμφωνία και αυτό επιβεβαιώνεται και στην ίδια συμφωνία δεν θα υπάρχουν πλέον παρκλήσεις. Όπως ξέρετε, στην Ιταλική πλευρά υπήρξαν πολύ μεγάλα εμπόδια, κυρίως λόγω προβλήματων που συναντήθηκα στην κλάδα της Σούζα. Και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, εγώ δεν έκανα σχόλια. Φυσικά από την πλευρά της Κομισιόν θα θέλαμε να είχαν προχωρήσει τα πράγματα γρηγορότερα. Αλλά όπως ξέρετε, τα μεγάλα σχέδια υποδομών αποτελούν την εξαίρεση παρά τον κανόνα. Πράγματι, το 2030 προβλέπεται τώρα ως ε, χρονοδιάγραμμα. Ξέρω ότι και από τις δύο πλευρές, και αν διαβάσετε τα ανακοινωθέντα τύπου του κυρίου Λάντ και του Πρωθυπουργού Λέτα, φαίνεται ότι αυτές αποτελούν τις ε, κύριες περιοχές προτεραιότητας ένθεν και ένθεν των συνόρων. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι εγώ να κάνω την δουλειά μου όσο πιο ενεργητικά μπορώ και ε, ελπίζω ότι οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να δώσετε και στον ε, διαδοχό μου θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Για την ερώτηση τώρα του κυρίου Ρικέ, η οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε θεωρείται ότι θα δινόταν για το διασυνοριακό τμήμα. Ένα τμήμα ε, της συμφωνίας ε, ήταν ότι και από την Ιταλική πλευρά θα υπήρχε μια κάποια καθυστέρηση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στη Σύραγα, αλλά όχι τόσο γρήγορα και όχι τόσο πλήρω όσο είχε προβλεφθεί. Τώρα, εγώ τι να σας πω, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει μέχρι το 2030, δεν μπορώ να μιλήσω για την Κομισιόν συνολικά και τώρα εν τω μεταξύ όσο ε, προχωρούμε με το έργο ε, δεν ε, θα υπάρχει ίσως και τόσο πολύ μεγάλη πίεση και πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει και στην περίπτωση Ισπανίας Γαλλίας και στα Ισπανικά σύνορα. Ναι, φυσικά, τα χρήματα είναι το παν. Και το κοινοβούλιο το γνωρίζει πολύ περισσότερο, γιατί τώρα έχετε εγκρίνει ένα προπολογισμό χαμηλότερο για πρώτη φορά από ό,τι στο παρελθόν. Όμως εδώ βρισκόμαστε. Εγώ κατανοώ το πρόβλημά σας και κατανοώ τα σχόλιά σας, αλλά τι να σας πω τώρα, δεν ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι όταν λείπουν τα χρήματα. Και για το λιμάνι στη Σλοβενία, για αρκετό καιρό δεν υπήρχε πρόβλημα γιατί για τη Σλοβενία είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σύνδεση με την κόπα και την πρόσβαση στη Μεσόγειο. Όμως είναι ένα ξεχωριστό τμήμα ε, έχουμε και το λιμάνι της Τεριέστης ε, εκεί κοντά. Όμως υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. νέα συμφωνία μεταξύ Ιταλών και Σλοβαίνων για μια κοινή υποδομή σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος δισταγμός που έχει αφαιρεθεί και από τα δύο μέρη. Και κάτι πολύ πιο σημαντικό και ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, πως υπάρχει τώρα ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ε, μεγάλα ιταλικά ε, λιμάνια στο βορρά, όπως είναι η Τραγέστη και η Βενετή, να συνεργαστούν περισσότερο με την κόπα. Και νομίζω ότι όλο αυτό προσθέτει μια ευρύτερη διάσταση Νομίζω το όραμα είναι σημαντικό και τώρα πιθανότατα το βόρειο τμήμα της ε, Μεσογείου στην Αδριατική θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι στο παρελθόν για να ανταγωνιστεί και με κάποιο τρόπο με την ε, δυτική πλευρά, με τα λιμάνια εκεί. Έτσι, λοιπόν, εγώ νομίζω ότι τα τελευταία 7 έτη έχουμε σημαντικές εξελίξεις, υπάρχουν ε, καλά σημάδια συνεργασίας, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει και το δικό σας κοινοβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπριχώση. για την έκθεση. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους για τις εκθέσεις και για την υποστήριξη που εξασφαλίζουν από την Επιτροπή. Και θα δούμε βεβαίω. και εάν μετά τις Αυτή με την προσοχή της Συνθεσή Επιτροπή των Μεταφορών θα δείχνει την ίδια επιμέλεια και το ενδιαφέρον, όπως και η προηγούμενη, από τον κύριο Παύλο Κώστα. Άλλωστε. Πολύ σωστά. Μιλήσατε για την Βόρεια Αδριατική. Ο Παύλο Κώστα ιδιαίτερα είχε ασχοληθεί με τη Βενετία. Σε ευχαριστώ λοιπόν όλους. Και προχωρώ στο επόμενο θέμα. Είναι μια ευχάριστη σύνδεση με το θέμα των λιμανιών. Αφήνω τους συντονιστές να αποχωρήσουν για να προχωρήσουμε την έκθεση του κ. Φλέκινστάιν. Thank you, Chairman. Can you just hang on a second till we... Δύο λεπτάκια αν θες να περιμένεις για να εκενωθεί η αίθουσα. Okay, Mr. Fleckenstein. Ports Ελάτε. Λιμενικές υπηρεσίε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρόταση τη Επιτροπή επικεντρώνεται σε τέσσερι κύριου τομεί Πρόσβαση στην αγορά, στις λιμενικέ υπηρεσίες, ε, η οικονομική διαφάνεια και συμβουλευτικά ή εποπτικά όργανα. Μετά από τις δύο πρώτες αποτυχίες πιστεύω ότι διδάχτηκε το δοχμά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναβαθμίσει την πρόταση. Αντίθετα, με, το, με τα πακέτα 1-2 περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα των ε, επιβατών και βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει κοινωνικός διάλογος. Υπάρχουν, ωστόσο, επικρίσεις Αρκετοί ήταν οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι διατυπώνουν αντιρρήσει ω προς τη διαφάνεια στην αλυσίδα των υποδομών και για τις αρχές εποπτείας. Το κείμενο της Επιτροπής μπορεί να τροποποιηθεί κατά τρόπο ώστε να οδηγήσει σε ε, καλώς τα λιμάνια χωρίς επιπλέον ε, προσκόμματα αλλά με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Η προσθέμενη αξία που ζητούμε πάντα είναι να περνάει μέσα από την ενίσχυση αυτονομίας ε, των λιμένων υποδομές παραδείγματι αυτόνομες ε, που δεν θα διοικούνται από ένα μακρινό Υπουργείο στην κυβέρνηση. Τα λιμάνια μπορούν να γίνουν ένα πραγματικό εργαλείο για την ε, ε, για την διατύπωση και ανάπτυξη μιας στρατηγικής επιχειρηματικής για την καλή λειτουργία της αγοράς και της εσωτερικής αγοράς. Και έτσι νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και ένα level playing field, ένα ισότιμο πεδίο αναμέτρησης. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίως πρέπει να εξεταστεί εκ παραλλήλου με δύο άλλες ε, προτάσεις. Καταρχάς, τη σχετική με την ε, με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εγκάρσιες κρατικές ενισχύσεις που αναμένουμε την επόμενη χρονιά και η οδηγία, την οδηγία για τις εκχωρήσεις που δεν έχει εγκριθεί. Και νομίζω ότι όσο δεν έχει ρυθμιστεί αυτό το θέμα των εκχωρήσεων δεν μπορεί να προχωρήσει συμφωνία ε, το θέμα αυτό. Για την ίδια τώρα την πρόταση. Είναι 84 τροπολογίες που έχω καταθέσει εγώ δεν αρκούν, όπως θα διαπιστώσουμε, αλλά βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή των συζητήσεων. Η μήνυα ακρόαση, αλλά και οι συζητήσεις με, με τα συνδικαλιστικά σωματεία και τους εκπροσώπους τους θα φέρουν, πιστεύω, και άλλες τροπολογίες. Η γενική προσέγγιση πέραν της ενίσχυσης αυτονομίας των λιμένων ε, δημιουργία μιας, ε, προβλέπει και τη δημιουργία μιας ε, υπηρεσίας υποβολής παραπώνων χωρίς επιπλέον όμως γραφειοκρατική επιβάρυνση και αυτό ισχύει και για τις διαβουλεύσεις με τους χρήστες των λιμένων που πάλι δεν θα πρέπει να οδηγήσει πλέον γραφειοκρατική επιβάρυνση. Ενώ και από αυτά που μας, λένε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκφραστούν στο διατακτικό με ουσιαστικό τρόπο, ε, να μην μείνουμε δηλαδή σε γενικόλογες τοποθετήσει, και δεν μπορούμε να έχουμε one size fits all. Πρέπει κάθε περίπτωση να εξετάζεται ε, ε, σωστά. Ε, επίσης, πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το πεδίο εφαρμογής. Η φθοκόρηση δεν έχει θέση εδώ. Γιατί αφορά ε, τις ε, υποδομές των λιμένων. Οι δε ε, υπηρεσίες ρημούλκησης θα πρέπει να εξεταστούν γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την ε, ασφάλεια στους λιμένες και άρα πρέπει και να υπάγονται στις ρυθμίσεις περί αλλά και να εξαιρεθούν από τη γενική ρύθμιση για την ε, ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά ακριβώς επειδή έχουν να κάνουν την ασφάλεια. Θα γίνουν σχετικές τροπολογίες. Ο αριθμός των ε, παρόχων και ο περιορισμός αυτού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιες αιτιολογίες που δεν αρκούν όμως. Νομίζω υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να περιορίζεται, ο αριθμός των παρόχων και το μέγεθος, η έκταση, η, ε, απλή, το απλό δυναμικό ενός λιμένα, δηλαδή πόσα πλοία μπορεί να χωρέσουν ταυτόχρονα. Ε, δεν έχει νόημα να έχουμε έναν πάροχο ο οποίο θα προσφέρει την υπηρεσία του ενώ κάποιο άλλο περιμένει στην ώρα για να πάρει σειρά. Η διαδικασία για την ε, εκτός θα πρέπει να προχωρήσει σε περίπτωση όπου η οδηγία για τις εκχωρήσεις οδηγεί σε προβλήματα. Εάν δηλαδή έχουμε περιπλοκή στους, ε, ως προς τη γραφειοκρατική επιβάρυνση, θα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Αυτό που δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση, αλλά έχει πιστεύω ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει να το επεξεργαστούμε περαιτέρω, θα είναι το cherry picking, η επιλεκτική δηλαδή, ε, η επιλεκτική ανάθεση να αποφεύγεται. Αυτό νομίζω όμως ήδη είναι ξεκάθαρο. Και τέταρτο σημείο, ο λιμένας θα πρέπει να είναι σε θέση να πληρεί τις προδιαγραφές του δεύτερου κεφαλαίου, τις ε, υπηρεσίες δηλαδή, και όχι με το PSO όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πέμπτο σημείο, η, τα τέλη, οι αποζημιώσεις για τις υποδομές θα πρέπει να έχουν τη σχετική κάλυψη ευελιμένε, εφόσον όμως τα κριτήρια, η κάλυψη, οι υποδομές είναι διαφανείς για τον ορισμό των τελών και πρέπει να είναι σε θέση. Θερυπή να προσφέρουν και εκπτώσεις ε, για να προωθήσουν μια στρατηγική ε, προώθηση ή για να προωθήσουν την περιφερειακή παραγωγή ενδεχομένως. Θα πρέπει να υπάρξει προσδιορισμός για το ύψος, ανάλογα βέβαια και με την ε, περιβαλλοντική διάσταση, αλλά και το μέγεθος ή το είδος των, ε, ε, των εκπτώσεων. Διαβουλεύσεις με τους λιμένες. Ήδη έχουμε με τους πλοηγούς ξεκινήσει διαβουλεύσεις και συγγνώμη, με τους χρήστες των λιμιών ξεκινήσει διαβουλεύσεις, αλλά θα πρέπει κάθε χρήστης να έχει τη δυνατότητα και να ενημερωθεί και να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Οι ε, χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση και να ενημερώνονται για την δομή των τελών και τα κριτήρια που έχουν επιλογή για αυτά. Και η διαβούλευση αυτή θα συζητήσει βεβαίως διάφορα θέματα, αλλά όχι το τελικό ύψο των τελών, γιατί αυτό είναι ένα ατομικό ζήτημα. Η αρχή εποπτείας, 7ο Θα είναι καταρχά μια γραμμή, μια, θέση, μια υπηρεσία υποβολή παραπώνων. Και έτσι, είτε πρόκειται για περιφερειακά δικαστήρια, είτε πρόκειται για ε, δικαστήρια ε, ανταγωνισμού, είτε για άλλες τοπικές αρχές εποπτείας, η δουλειά που θα κάνει θα πρέπει να είναι ουσιαστικά η ανεξάρτητη εποπτεία, χωρίς όμως να υπαγορεύουν αυτές οι αρχές εποπτείας, πώς θα γίνεται η οργάνωση του λεμένα. Και θα πρέπει να γίνεται, ε, να ορίζεται ποια είναι αυτή η υπηρεσία παραπώνων, χωρίς όμως να δημιουργούνται νέες δομές. Και αυτό σημαίνει όχι, όχι την υποβολή γενικώ ε, παραπώνων, αλλά την υποβολή συγκεκριμένων προσφυγών με βάση το ισχύον ε, δίκαιο. Και βέβαια πρέπει να μεριμνάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τήρηση του κανονισμού δεν υπάρχει τέτοια είδου υπηρεσία εποπτεία ε, σε κάποια χώρα θα πρέπει να δημιουργηθεί ασφαλώ. αλλά εάν σε άλλες χώρε υπάρχει δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί κάτι καινούριο. 3 Δεκεμβρίου προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Δύο, και, 2 ή 3 ε, συνεδριάσεις και οδών Για τις 12 Δεκεμβρίου προβλέπω την πρώτη 11 Φεβρουαρίου κατά πάσα πιθανότητα ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και Μάρτιο του 2014 στη Σύνοδο την ψηφοφορία. Πρώτες αντιδράσεις εκτός του Κοινοβουλίου από ΦΥΠΟΡΤ, ΕΣΠΟ είναι σχετικά θετικές. Με τα συνδικάτα είμαι σε επικοινωνία, υπάρχουν κάποιες ε, επιφυλάξεις επί της ουσίας. Και έτσι πρέπει να πω ότι τίποτα δεν έχει κλείσει όσο δεν έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Αυτά και περιμένω την καλή συνεργασία με τους συναδέλφους. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κομουτσάκος, Σεμπάκα, Ράντα, Ρίλς, ο Σχιώδης. Τέσσερα λεπτά γι' αυτό και μετά Ρίκε, Μαντάλεν, Φεντάντζα, Α, και η κυρία Γιάλα Τέσσερα λεπτά για τους κοιόδης, δύο λεπτά για τα μέλη. Εντάξει, βάζω το ρολό γιατί αλλιώς χανόμαστε. Κύριος Κουμτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναλαμβάνουμε και ξεκινάμε τη συζήτηση ενός ε, πολύπλοκου ε, ζητήματος και η ελπίδα όλων είναι ε, αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε. Ε, δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε από το βαρύ παρελθόν, δύο αποτυχημένων προσπαθειών, ε, αλλά με αποφασιστικότητα και ευελιξία κυρίως και επικοδομητικό πνεύμα να επιχειρήσουμε και να καταφέρουμε αυτή τη φορά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς πιστεύω αυτά, θέλω να καλωσορίσω την ε, παρουσίαση και την προσπάθεια που έχει κάνει ο εισηγητής, ο συνάδελφος κ. Φλάκενστάιν. Το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεών του κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω όμως ότι ταυτόχρονα θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε ε, διάφορα σημεία τα οποία χρειάζονται ίσως κάποια διευκρίνηση ή ορισμένες τροπολογίες. Αλλά αυτό το οποίο κυρίως θέλω να συγκρατηθεί είναι ότι η δουλειά ε, που έχει κάνει και που μας παρουσιάζει σήμερα σαφώς κινείται στη σωστή κατεύθυνση και την καλωσορίζω. Ξεκινάω με το θέμα της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής. Ε, συμφωνώ απολύτως με την προσέγγιση του και την αντικατάσταση, αν θέλετε, της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής από την έννοια και την ανάγκη να υπάρχει γενικώ μια ανεξάρτητη εποπτεία, χωρίς να δημιουργούμε μια νέα δομή. Ε, αυτό το οποίο όμως πρέπει να, να διασφαλιστεί ότι όποιος φορέας διαμορφωθεί πρέπει να λειτουργεί <clears throat> ανεξάρτητα. Ε, όσον αφορά ε, στην, διαγραφή του άρθρου 18 που αφορά στη συνεργασία ε, μεταξύ ανεξάρτητων εποπτικών αρχών γενικά συμφωνώ με την διαγραφή όλων των επιμέρους υποχρεώσεων ταυτόχρονα όμως θα μπορούσε κάποιος να εξετάσει τη δυνατότητα κάποιας πλατφόρμας διαλόγου, πολύ ευέλικτης, για την ανταλλαγή πληροφοριών και των πρακτικών. Αλλά γενικά συμφωνώ με την διαγραφή ε, του άρθρου 18. Τώρα, όσον αφορά τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων ε, υπηρεσιών του άρθρου 6 ε, και εκεί πιστεύω ότι είναι σωστό ότι <coughs> εντάσσονται ε, ακόμα ε, τρία κριτήρια ε, που θα μπορούν να δικαιολογούν τον περιορισμό των παρόχων είναι η, ο μικρός χώρος από πλευράς θαλάσσης, το μέγεθος, το μικρό μέγεθος του λιμένα και η μειωμένη παραγωγική ικανότητα και βεβαίως η ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας προστασίας του περιβάλλοντος και τα τρία αυτά κριτήρια νομίζω ότι συνενούν στο να έχουμε μια ε, περιορισμένο αριθμό παρόχων όταν αυτά, αυτές οι τρεις προϋποθέσεις συνυπάρχουν. Ε, όσον αφορά την, ε, την διαβούλευση με τους χρήστες ε, του Λιμένα, υποστηρίζουμε την τροπολογία και την ιδέα του κυρίου Φλάνκενστάιν. Τώρα, όσον αφορά την ανάγκη της αυτονομίας του διαχειριστικού φορέα, του λιμένα, ε, πιστεύουμε ότι ο συγητής κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ε, πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την οικονομική στρατηγική του, ε, τηρώντας βέβαια κάποιες βασικές αρχές. Η διαφάνεια είναι απαραίτητη κυρίως εκεί που έχουμε περιπτώσεις κρατικής βοήθειας. Τέλος, ε, όσον αφορά την έναρξη, ε, δώστε μου ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την έναρξη ισχύω του κανονισμού, ε, πιστεύουμε και εμείς ότι μπορεί να ξεκινήσει μίνιμουμ δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση εφημερίδας και κυβερνήσεως. υπάρχουν δύο σημεία, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε αν έφυγα από τον χρόνο, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία είναι σημαντικά. Το dredging, ε, συμφωνούμε με την διαγραφή, αντιλαμβανόμαστε τη λογική του, του εισηγητή, όμως θα πρέπει να εξετάσουμε και μια διάσταση του dredging που είναι ιδιαίτερη και πρέπει να μας απασχολήσει. Και αυτό είναι ότι αρκετές φορές το dredging εμέσως αλλά σαφώς παίρνει μορφή κρυφής κρατικής ενίσχυσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε. Okay. Ε, και για το πιλοτάζ πρέπει να βρούμε μια νέα ισορροπία μεταξύ της πλήρους διαγραφής και του κειμένου που έχει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεμπάκερ, παρακαλώ μείνετε στα τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στα Ολλανδικά λέμε τρίτη και τυχερή. Ελπίζω αυτό να συμβεί και με αυτή την ε, πρόταση. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν ήταν για μας ε, ήδη στη σωστή κατεύθυνση κινούταν, αλλά και τώρα ε, υπάρχουν νέες προσθήκες που ενισχύουν την αρχική πρόταση. Πρέπει όμως να δώσουμε έμφαση στη διάκριση μεταξύ των διαφόρων λιμένων, ανάλογα με το μέγεθος και το καθεξής. Όμως θα πρέπει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε κάποιες γενικές ε, συμφωνίες μέσω αυτού του κανονισμού. Δεν συμφωνώ με την προσαρμογή του πεδίου εφαρμογή που προτείνει ο εισηγητής. Βεβαίως ω όσο πάντα και τώρα θεωρούσα ότι πρέπει να ε, υπάρχει μια ανοιχτή προσέγγιση ό,τι αφορά τι εξουσίε. Μπορούμε έτσι να έχουμε καλύτερη παροχή υπηρεσιών και να αυξηθεί και ο ανταγωνισμό. Όχι μόνο δηλαδή να αυξηθεί ο ανταγωνισμό μεταξύ των λιμένων, αλλά να βελτιωθεί και να έχουμε τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία ε, και τον καλύτερο δυνατό ανταγωνισμό και στο ιστορικό των λιμένων. Και αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί. Επομένω, πλέον ε, Πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω το πεδίο εφαρμογή. Ε, θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια καλύτερη δέσμη από ότι ε, η υφιστάμενη πρόταση του εισηγητή. Ε, επιπλέον δεν είμαστε υπέρ των, του επιπλέον διοικητικού άχθου και των διοικητικού κόστου. Και εδώ είναι σημαντικό το ζήτημα και της επίβλεψη. Εδώ πέρα μπορεί να υπάρξει κατάλληλη συμφιλίωση και η προσέγγιση του εισηγητή σίγουρα χρήση, στήριξη στην οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω. Για τους χρήστες ε, του λιμένα θεωρούμε και πάλι ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά τις ε, επιπλέον εμπορικές ε, ελευθερίες που μπορούν να δεθούν με τον προσδιορισμό κάποιων τελών πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα εχέγγυα βεβαίως, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Δεν ε, συμφωνούμε με τη συζήτηση από τη μετάβαση μια σύμβαση από τη μία επιχείρηση στην άλλη ε, να ε, έχουμε πολύ αυστηρές προδιαγραφές για το προσωπικό. Αυτό είναι ζήτημα του κράτους μέλους, αρμοδιότητα του κράτους μέλους, με διαφορετικά καθεστώτα σε ό,τι αφορά ε, το προσωπικό και όλη αυτή η συζήτηση των κοινωνικών υποθέσεων θα πρέπει να περνάει από μια κοινωνική συζήτηση, κοινωνικό διάλογο. Κάποιες τροπολογίες ε, στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δίνουμε ώστε να τον περισσότερες δυνατότητες για τον κοινωνικό διάλογο τα πάντα πρέπει να τίθενται επιτάπητο και δεν θα ε, οδηγηθούμε έτσι στο, στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ημερομηνίε. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια ε, αναβολή για δύο-τρία χρόνια, γιατί έτσι ε, υπάρχουν καθυστερήσεις, πρέπει να τα κλείσουμε αυτά πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός, με κατάλληλο πεδίο εφαρμογής, έτσι μόνο καλύτερα θα είναι η θέση των λιμένων μας. Και έτσι θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να έχουμε ένα κατάλληλο ε, πακέτο, μια δέσμη μέτρων για τους λιμένες. Ευχαριστώ, Bradburn, για τέσσερα λεπτά. Ούτε καν τέσσερα λεπτά δεν θα μιλήσω, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για ε, το έργο του σίγουρα πρόκειται για σαφή βελτίωση σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Συμφωνώ ιδιαίτερως με αυτή την πρόταση για το ανεξάρτητο εποπτικό φορέα. Έτσι θα αποφύγουμε αυτή την ε, περίτη γραφειοκρατία. Όμως έχω κάποια σημεία επιφύλαξης δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση, παρότι έχει τροποποιηθεί καταλήλω. Είναι η τρίτη, πρόταση, τρίτη φορά που μια τέτοια πρόταση έχει ε, υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και δύο φορές έχει απορριφθεί και πολύ σωστά απορριφθεί. Ε, Κάποιε φορέ αναρωτιέμαι τι ακριβώ δεν κατανοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω και να έχει, η πρόταση είναι εξαιρετικά γραφειοκρατική και παρεμβατική, θεωρώ. Δεν αναγνωρίζει την ανάγκη των αγορών να λειτουργούν ελεύθερα και τις διαφορετικές ανάγκες ε, των ε, λιμένων ε, που λαμβάνουν δυτική χρηματοδότηση σε σχέση με με τους λιμένες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά και, το, και τους όρους του, ανταγωνισμού, επειδή έχουμε όλο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, δεν χρειάζεται να υπάρξει κανονισμός. Σίγουρα όχι αυτή τη χρονική στιγμή πρέπει να δούμε τι θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική της για τις κρατικές ενισχύσεις ε, και επιχορηγήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ξέρετε Πρόεδρε, έχουμε ιδιαίτερα ε, επιτυχημένο ιδιωτικό τομέα στους λιμένες και έτσι πλέον ε, ε, τίθεται σε κίνδυνο ε, μεγάλος αριθμός θέσεων εργασία, αλλά και λειτουργία του των κλάδου των λιμένων. Δεν υπάρχει μία λύση για όλους, one size fits all. Γι' αυτό, Πρόεδρε, συμπερασματικά, εγώ θα υποβάλω τροπολογία να απορριφθεί η πρόταση. Και ελπίζω στην εξέταση αυτών των συντημάτων ε, να καταλήξουμε στην απόρριψε τις πρότασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία. Η για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ τάσουμε κατά των προτάσεων και μετά ακόμη τις ε, προτάσεις του εισηγητή καλύπτεται κατά 80% το ποσό των χρηστών από τις υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας των λιμένων. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να εισαχθεί νέα νομοθεσία. Είμαι βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ότι θα περάσει αυτό και μετά θα έρθουμε ένα τέταρτο πακέτο για τους λιμένες ώστε να ε, καταστήσει παροχημένο και το τρίτο πακέτο. Ο κανονισμός δεν είναι η κατάλληλη μορφή για την αντιμετώπιση των διαφόρων ε, συνθήκων που επικρατούν στους ευρωπαϊκούς λιμένες σε διαφορετικές χώρες και περιοχές, έχοντας δε ε, συνεργαστεί με την, έχοντας ακούσει τη γνώμη των, ε, ε της των Λιμένων Βορείου Γερμανίας, πάλι βλέπω ότι και αυτοί διαφωνούν, πρόβλημα είναι και η βυθοκόρηση και η πλοήγηση. Ξέρω ότι βεβαίως μεριμνά ο εισηγητή, αλλά δεν νομίζω ότι η Επιτροπή θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις, ε, την ανάγκη να, να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογή. Ακόμα δε και αν αποκλειστούν οι πλοηγοί από το πεδίο εφαρμογή, κανεί δεν μα λέει ότι από την ώρα που θα αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα δεν θα ανοίξουν πόρτα και παράθυρα για να μπουν, από την, ε, για, για να μπουν τελικά στο πεδίο εφαρμογή. Επίσης συμφωνώ με το Συνδικάτο των Ευρωπαίων Λίμεν Εργατών που τάσσονται κατά της απαγόρευσης ε, της ε, απεργίας ή του περιορισμού του δικαιώματος στην απεργία γιατί ξέρετε ότι υπάρχει ε, μια σχετική πρόταση που θα πρέπει να διαγραφεί απολύτως εάν πρόκειται τελικά να επεξεργαστούμε την ε, πρόταση του κανονισμού, αν δεν απορριφθεί δηλαδή εξ αρχής. Με λυπείται ότι ο κύριος Φλέκενστάιν δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Υπήρξε μια προσπάθεια αντίστοιχα για τον περιορισμό της, ε, του δικαιώματο στην απεργία με το σιδηροδρομικό πακέτο και τώρα βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέρχεται με τις προθέσεις που είχε διατυπώσει ήδη από τη δεύτερη Επιτροπή Μόντι για περιορισμό λοιπόν του δικαιώματος της απεργίας και στα λιμάνια. Η ΕΤΕΦ, Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμενατεργατών, ε, πιστεύει όπως και εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει πρώτα το κάρο και πίσω τα βόδια ε, γιατί δεν έχει ακόμα προχωρήσει την οθέτηση της οδηγίας για την, για την εκχώρηση, ένα κείμενο το οποίο δεν έχει καν ε, εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και άρα δεν μπορεί να ε, αποτελέσει δεσμευτικό έγγραφο αυτός ο κανονισμός, εάν και εφόσον προχωρήσει. Το άρθρο 18.1 αναφέρεται σε μια δομή, σε ένα δίκτυο το οποίο ε, θα πρέπει να επανεξεταστεί με πολύ μεγάλη προσοχή. Η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, δεδομένης και της όλης συζήτηση για, την, ε, για το σκάνδαλο NSA θα πρέπει να κρυθεί τουλάχιστον ανεπαρκής. Ευχαριστώ πολύ. Η λυπή συνάδελφη, δύο λεπτά έκαστος ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι οι οδηγίες για τους λιμένες είναι αρκετά φαρδιές φαίνεται γιατί τις πλένουν, τις ξεπλένουν και πάλι αρκετά φαρδιές είναι. Και φαρδιές μένα αλλά μπαίνουν σιγά σιγά στο πλήσιμο, παραμένουν όμω φαρδιές όπω πούμε. Τις απορρίπτουν λοιπόν τα δύο άκρα του κοινοβουλίου. Ίσως εάν ξαναμπούν λίγο ακόμα και πανεστιάσουμε τις ε, προτάσεις να εγκριθούν. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις αναφερθήκατε σε πλοήγηση ή σε ρημούλκηση τελικά. Γιατί εγώ από την έκθεση σας φαντάστηκα ότι για πλοήγηση θα έπρεπε να μιλάτε και όχι για ρημούλκηση. Πάντως είναι ούτως ή άλλως ε, το, τα, από τα πιο σημαντικά θέματα για την ασφάλεια των λιμένων. Η πλοήγηση θα πρέπει να αποκλειστεί ασφαλώς. Αλλά ίσως και η ρημούλκηση για τους ίδιους λόγους. Και η πρόσδεση. Το ίδιο και για τη βυθοκόρηση που αφορά υποδομές. Βέβαια, αν αποκλείσουν τα πάντα, θα μείνει και πολύ ουσία στην πρόταση. Η δεύτερη παρατήρηση που έκανε η προηγούμενη ομιλήτρια είναι η εξή. Ότι όσο δεν υπάρχει αυτή η οδηγία για τι εκχωρήσει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί παραμένουν ε, αμφιβολίες ως προς την εξέλιξη, την ζωή μετά την έκθεση αυτού του κειμένου. Και επίσης η αρχή εποπτείας είναι απαραίτητη. Βεβαίως βλέπω ότι θέλετε να αξιοποιήσετε οι υφιστάμενες δομές και αρχές για να αποφευχθεί η γραφειοκρατία. Αλλά θα είναι πολύ διαφορετικές οι λειτουργίες αυτών των αρχών εποπτείας, ανακράτος μέλος, θα είναι πολύ αφήσει ακόμη και η εικόνα που θα έχει ο χρήστη του λιμένος για το τι μπορεί να περιμένει. Και αυτό ίσως ε, θα ήταν επιβλαβές. Προτιμώ να παραμείνει η πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ, Βαντάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν περιμένω αυτή την πρόταση, γιατί σε ό,τι αφορά τι ε, κρατικέ ενισχύσει στου λιμένε. Πρέπει να περιμένουμε τι προτάσει που θα έρθουν από πλευρά ε, κομισιών ακριβώ για τι κρατικέ ενισχύσει. Επομένω, ε, αν ζυγίσουμε λίγο τι δύο προτάσεις, τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Το πιο σημαντικό είναι το τρίτο, τρίτο συγγνώμη, κεφάλαιο για την διαφάνεια και την αυτονομία. Όμως ε, με ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο έχει ε, διαμορφωθεί αυτή η πρόταση. Έχουμε ένα πολύ γραφειοκρατικό σύνολο. Επομένως είμαι ιδιαίτερα επικριτικός ε, απέναντι σε αυτή την πρόταση και επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε έναν ολόκληρο κοινωνικό διάλογο με κοινωνικές διατάξεις, ελάχιστες απαιτήσει, όπως έχουμε δει συχνά και στην αεροπορία το δάμε αυτό, ε, και πραγματικά δεν χρειαζόμαστε τέτοιε συζητήσει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η βασική μου παρατήρηση, Πρόεδρε. Η δεύτερη αφορά το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Ο εισηγητή ε, δικαίω μιλά ε, για την ασφάλεια. Δυστυχώς ξεχνάμε ότι για την ασφάλεια είναι σημαντικές και υπηρεσίες πρόσδεσης ε, των πλοίων στο λιμένα ε, που διασφαλίζουν ότι δεν θα φύγει το πλοίο από το λιμάνι. Επομένω, ε, και εδώ είναι σημαντικό και θα πρέπει να υπάρχει σαφής εξαίρεσή τους από τον κανονισμό. Μετά, στο άρθρο 14 θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην έννοια του πράσινου λιμένα, να συμπεριλάβουμε και την οικολογική διάσταση για ε, αυτό το κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πραγματικά έχω προβληματιστεί πάρα πολύ για αυτή την πρόταση κανονισμού και γιατί φτάνει αργά, καθυστερημένα. Δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας πριν το τέλος της θητείας. Επίσης, είναι αποδυναμωμένη από τα πλέον θεμελιώδη στοιχεία που ήταν αυτά τα οποία στο παρελθόν ήταν σημαντικά, δηλαδή υπηρεσίε για τους επιβάτες και για τα εμπερεύματα. Υπάρχει βέβαια και ένα θετικό στοιχείο για την υπογράμμιση και ο συγητής που αφορά το θέμα της ε, χρηματοοικονομικής διαφάνειας ε, και κατόπιν γίνεται λόγος για απελευθέρωση ορισμένων λιμενικών υπηρεσιών που κατά την άποψή μου δεν είναι και ιδιαίτερα σημαντικές αυτή τη στιγμή. Έχουν χαμηλό αντίκτυπο προς το κόστος. Όλες οι έρευνες μας λένε ότι ένας εμπορικός σε ένας επιχειρηματίας δεν επιλέγει ένα λιμάνι βάσει αυτών των υπηρεσιών αλλά βάσει άλλων στοιχείων και επίσης για το θέμα της πλοήγησης αλλά και για το θέμα της ε, ρημούλκησης ε, και αυτά είναι στοιχεία που σχετίζονται πολύ στενά με τις απαιτήσει ασφάλειας. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει και τόσο μεγάλη διαφορά γιατί αν ένα πλοίο βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση κοντά σε ένα λιμένα και το πρώτο που ενδιαφέρει ε, είναι η ρημούλκηση για να σωθεί αυτό το σκάφος και κατόπιν η πλοήγηση. Έτσι λοιπόν αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη βέβαια. Λέμε ότι αν αφαιρέσουμε τη βυθοκόρηση όπως θέλει ο συγητής, και εγώ συμφωνώ, αν αφαιρέσουμε και την πλοήγηση όπως θέλει ο συγητής, και πάλι συμφωνώ και εγώ θα έλεγα να αφαιρέσουμε και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, δεν μένει τίποτα. Αλήθεια είναι. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση συγκρονισμού δεν θα έπρεπε να γίνει από αυτού του όρου και ίσω θα ήταν καλύτερο να σκεφτούμε μια οδηγία παρακανονισμού. Παρακαλώ, κύριο Τικράνη. Ευχαριστώ. Εγώ θυμήθηκα ε, το δυσάρεστο βίωμα που είχαμε με τον εκβιασμό και στο Στρασβούργο και θα θυμάστε κύριε Σίμψον και κατόπιν η Κομισιόν καθυστέρησε πέντε χρόνια για να καταθέσει μια νέα πρόταση και τη φέρνει στο τέλος της αιτίας μας. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι και αρκετά τολμηρή η πρόταση και πραγματικά η βούληση είναι να μην ε, έχει επιτυχία. Εγώ νομίζω ότι είναι ε, προφανής η βιωσιμότητα της πρότασης αυτής ε, και έχουμε και το χρονικό ενός πρώην αγγελθέντους θανάτου, όπως ξέρετε. Είναι ένα μεγαλό λογοτεχνικό έργο και εγώ νομίζω ότι αυτό θα γίνει με αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Το 90% των εμπορευμάτων μας ε, εξάγονται μέσω των λιμένων ε, και είναι σημαντικοί λιμένες ε, προκειμένου να υπάρχουν συνέπειες σε όλη την ε, αλυσίδα. Υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, που θέλουν κάποια περαιτέρω προνόμια. Εγώ δεν θέλω τώρα να τα αναφέρω ε, αυτά. Μα θυμίζουν παλιές ταινίε. Όμως η πρόταση είναι πάρα πολύ ντροπαλή, δεν είναι καθόλου τολμηρή. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσε εξαιρέσεις και να μιλάμε για απελευθέρωση υπηρεσιών. Υπάρχουν κάποιες υπερβολές σε σχέση με την επιβολή τετλών λοιπόν για τα τέλη, με την υποβολή τελών για τις υποδομές. Εγώ συμφωνώ με τον συγητή όταν μας προτείνει ότι οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να παρέχουν σε αυτούς τους υπηρεσίες. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός ε, μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ πρέπει να έχουμε περιορισμό και κοινωνικό ντάμπινγκ όταν δεν χρειάζεται ε, να ε, θέτουμε πρόβλημα γιατί τα δικαιώματα των εργαζομένων νομίζω ότι είναι ήδη προστατευμένα από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Γιάλε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ έχω την εντύπωση ενός ε, ντεζαβί, δηλαδή σαν να ξαναβλέπω το ίδιο κείμενο και μάλιστα ακόμη και πιο περιορισμένη είναι αυτή η πρόταση που μας παρουσιάζει η Κομισιόν σήμερα, ακόμη πιο αποδυναμωμένη από τις δύο τελευταίες φορές. Και εμείς ε, εδώ τι κάνουμε τελικά, μειώνουμε κάθε φορά, περιορίζουμε κάθε φορά το παιδί εφαρμογής ώστε να περάσει τελικά. Εγώ πραγματικά αναγνωρίζω τη δουλειά του εισηγητή, όμως δεν μπορώ να καταλάβω τελικά ποιος θα εφαρμόσει το νόμο. Αν ε, εδώ προσπαθούμε τελικά να έχουμε καλύτερη νομοθέτηση και επίσης γιατί να έχουμε ένα κανονισμό δηλαδή να έχουμε κανόνες ε, άμεσης εφαρμογής. Και όταν λείπουν διάφορα στοιχεία, βυθοκόρηση, ρημούλκηση κτλ. Σε ποιον θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Σε ποιον θα εφαρμοστεί η νομοθεσία. Εγώ καταλαβαίνω ε, βέβαια το πρόβλημα που τίθεται. Βέβαια δεν συμφωνώ 100% με τα συνδικάτα, αλλά ίσως ε, θα έπρεπε να συζητήσουμε μαζί τους ε, για να αποφύγουμε να ξεσπάσουν κάποιες απεργίες. Και πρέπει να τα καταφέρουμε καλά αυτή τη φορά, όχι όπως κάναμε για το handling στις αεροπορικές υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τώρα τις εθνικές ενισχύσεις. Είπαμε ότι θέλουμε διαφάνεια. Όμως ούτε δεν το πετυχαίνουμε εδώ. Επομένως δεν καταλαβαίνω ποια είναι η χρησιμότητα της πρότασης και το ίδιο, το ίδιο ισχύει με την ομοσπονδιακή δομή γιατί εμείς έχουμε ένα δίκτυο λιμένο στην Ισπανία που είναι αυτόνομα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορούσαμε να το εντάξουμε αυτό το στοιχείο και υπάρχουν και άλλα θέματα όπως είναι η συνεργασία, το θέμα ε, τη σύνδεση με τις πόλεις. Αυτά τα θέματα δεν εμφανίζονται καθόλου και δεν ξέρω αν θα είμαστε κανεί να τα εντάξουμε στην πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να... Πριν ζητήσω από την Επιτροπή να λάβει το λόγο, θέλω και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εάν βγάλουμε την πλοήγηση, τη βυθοκόρηση, όλα αυτά τα θέματα για τα οποία και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να βγουν. Και αφού το handling φορτίου η Επιτροπή ίδια το βγάλε έξω. Δηλαδή ένα πακέτο για λιμάνια που δεν καλύπτει το, την, ε, τις υπηρεσίες εδάφους για το φορτίο και βγάζει και τη μυθοκόρηση και την, πλοιο, και όλα αυτά, ε, ρωτώ, μένει τίποτα μέσα, έχει κανένα λόγο να το συζητάμε όλο αυτό το πράγμα. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή. Και επίσης, ξέρω ότι έχει δουλέψει πολύ σκληρά ο εισηγητής, έχει δουλέψει σκληρά για να μπορέσει να δώσει κάποια ουσία σε αυτήν την πρόταση. Αλλά, από όσα λένε και οι συνάδελφοι, γιατί είναι ομόφωνη πιστεύω η εντύπωση ότι πάμε για μια τρίτη απόρριψη. Άρα σε άλλα τρία χρόνια περιμένουμε να δούμε μια νέα πρόταση από την Επιτροπή. Εμένα όμως αυτό που με ανησυχεί είναι το θέμα της αξιοπιστίας. Γιατί πριν πάει στο Συμβούλιο και <laughs> κύριος είδε τι θα πούνε και αυτοί από την πλευρά τους, για να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία μας θα πρέπει να μην προσπαθούμε να νομοθετούμε μόνο και μόνο για να νομοθετήσουμε. Γιατί, ναι, εάν είχαμε το φορτίο, το handling πολύ καλά, να το, να το πολεμήσουμε, θα γινόταν και καμιά αντίδραση έντονη κτλ. Το ζητήσουμε. Αλλά μπορεί και αυτό να είναι ο λόγο για τον οποίο ε, δεν έχει μπει το φορτίο μέσα, γιατί ίσω θέλουν να αποφύγουν τι αντιδράσει. Ε, εάν όμω δεν μπορούμε να πείσουμε ότι πρέπει να μείνει το handling των φορτίων, εάν δεν μπορούμε να πείσουμε ότι πρέπει να μείνει η βυθοκόβευση, αν δεν μπορούμε να πείσουμε ότι πρέπει να μείνει η πλοήγηση, ε, τότε πώ είναι καλύτερα να αποσυρθεί η πρόταση. Παρακαλώ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μεγαλειώδης εισαγωγή σας. για την εισήγηση. Ε, θα ήθελα να πω, έχοντα ακούσει και τον συγητή και βέβαια αρκετού από του ε, βουλευτέ σα, ότι τόντι έχουμε τα σωστά συστατικά. Τα συστατικά που θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο δεν ε, θα αφορά μόνο το άνοιγμα των αγορών και Λυπάμαι. Ναι, δύο φορές έχουμε υποβάλει πρόταση. Δύο φορές ήταν προτάσεις όπου στόχος ήταν αποκλειστικά το άνοιγμα στον ανταγωνισμό των λιμενικών υπηρεσιών. Το πήραμε το μάθημα. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο δυστυχώς έρχεται με κάποια καθυστέρηση η πρόταση, αλλά να, έπρεπε να κάνουμε την ε, σοβαρή δουλειά, τις ευρείε κοινέ διαβουλεύσεις για να αντιληφθούμε και να μεταφράσουμε σε ένα νομικό κείμενο τι ουσιαστικέ παραμέτρους και της λογοδοσίας και της ασφάλειας δικαίου μπορείτε να μας επικρίνετε για πολλά πράγματα. Αλλά αν κοιτάξετε τις διάφορες πτυχές που καταγράφει το κείμενο, είμαι πεπισμένος ότι θα πιστείτε πως πρόκειται για στοιχεία που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν κάθε εμπλεκόμενο φορέα και βέβαια τις αρχές διαχείρισης λιμένων πρώτα απ' όλα, για περισσότερη λογοδοσία, για περισσότερη διαφάνεια, εν τέλει για λιμάνια πιο αποτελεσματικά, για λιμάνια πιο καλά εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πολλοί από εσά επανέλαβαν τη βασική αυτή ιδέα και τη σημασία των λιμένων και στις μεταφορές αλλά και στην οικονομία γενικότερα η πρόταση του εισηγητή είναι μια καλή προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση κάποιων πτυχών, όπου ίσως να το παρατραβήξαμε. Επί παραδείγματι, απλούστευση της προς και προς τη επιπλέον ευελιξία που αναφέρει ο κύριος Φλέκνισταϊν για τις υπηρεσίες, για την εποπτεία, που έχει συζητηθεί με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε πολλές από τις τροπολογίες του εισηγητής διατυπώνει με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση ακόμη την αρχή της αυτονομίας των λιμένων. Μία αρχή, μία από τις αρχές που και εσείς και εμείς ασφαλώς έχουμε ε, διεκδικήσει εδώ και χρόνια. Μια άλλη πτυχή και είναι πάλι θέμα διευκρίνησης πιστεύω για την πλοήγηση και τη βυθοκόρηση. Στόχος δεν είναι ο αποκλεισμό των δύο αυτών ε, βασικών υπηρεσιών από τα κείμενα, αλλά να ε, καταδειχθεί σαφώς ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για υπηρεσίες καλυπτόμενες αποκλειστικά από την αρχή της διαφάνειας, από το από το σύστημα διαφάνεια προτείνουμε και βέβαια δεχόμαστε έτσι τις τροπολογίες του εισηγητή διότι πιστεύουμε ότι οι δύο αυτές οι υπηρεσίες με άμεσο κόστος η μία και έμεσο η άλλη στον, για τον χρήστη είναι σημαντικό κομμάτι της όλης αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των λιμένων. Και η προσθεμένη αξία βεβαίως ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άλλες πτυχές σημαντικές για μας με τις τροπολογίες που προτείνετε κύριε Φλέκινστάιν. Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί προσπαθούμε καλύτερα να προσαρμόσουμε την έννοια των αποκλειστικών δικαιωμάτων και την χρήση αυτών. Και εδώ το κείμενο πρέπει να πω ότι είναι μια σημαντική νομοθεσία. Προσφέρει ασφαλεία δικαίου στο γεγονός ότι τα αποκλειστικά γεγονότα, ε, δικαιώματα μπορούν να χορηγηθούν σε μια σειρά από υπηρεσίες λιμένων ανάλογα με την προσέγγιση σε κάθε περίπτωση και σε κάθε χώρα. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε στην ε, απαρίθμηση παραπομπών στους υφισταμένους νόμους ε, παραδείγματι καθεστώς εκχωρήσεων και καθεστώς δημοσίων συμβάσεων, κρατικών συμβάσεων, ε, γιατί αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της ασφάλειας δικαίου. Ε, ομοίως, όταν μιλούμε για κοινή ταξινόμηση σκαφών και τη διάσταση του χρόνου για την τακτική ε, επικαιροποίηση με τις ε, κατεξουσιοδότης συμπράξεις ε, και η οικονομική και η υπευελοντική διάσταση θα λαμβάνονται υπόψη, διότι πιστεύω ότι αν πρόκειται να ληφθούν υπόψη, αν πρόκειται να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι επενδύσει για την αγορά ενός σκάφου, θα πρέπει και ο επενδυτή να έχει επαρκή ασφάλεια δικαίου για να γνωρίζει αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματα αυτά που θα έχει αγοράσει σε περισσότερου του ενό λιμένες. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά είναι πολύ διαφορετικό το κείμενο σε σχέση με αυτά τα οποία συζητήθηκαν στο παρελθόν. Με πολλούς από τους παρισταμένους ε, έχω γνώση του γεγονότος. Πιστεύω όμως το σχέδιο εκθέσεως είναι μια πολύ καλή βάση για να γίνει εξασφαλιστή πρόοδος. Ευχαριστώ. Κύριε Φλέκενστάιν, σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα. Σε κάποια λίγα σημεία για, για την πλοήγηση θα το συστήσουμε ε, στις λεπτομέρειες του. Η θέση ισχύ θα πρέπει να εξαρτηθεί παραδείγματι από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα έχει προχωρήσει ο κανονισμός. Για την οδηγία για τις ε, εκχωρήσεις είπα ότι θα πρέπει να ψηφιστεί αλλιώς δεν ε, έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Διαφορετικές δομές για τις ε, αρχές εποπτείας. Δεν σημαίνει για μένα ότι δεν μπορεί να υπάρξει επαλήθευση. Εκτός και αν δεν ξέρουν τι πρέπει να επαληθεύσουν. Είναι ξεκάθαρο όμως θα πρέπει να επαληθεύουν αυτές οι αρχές. Τώρα, ποια αρχή θα είναι, εάν θέλει ένα δικαστήριο ανταγωνισμού, εάν θα είναι μια αρχή εποπτείας, οτιδήποτε από το ένα κράτος στο άλλο, αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Εφόσον υπάρχουν τέτοιε αρχέ δεν χρειάζεται να εφεύρουμε νέε. Και τελευταία, η πρώτη τελευταία πρόταση, οδηγία ή κανονισμός. Ή θα βρούμε μια λογική λύση όπου θα πούμε ότι κάναμε μια σωστή δουλειά πλέον και έτσι μπορούμε και κανονισμό να έχουμε και οδηγία ή αλλιώς τα αφήνουμε όλα ε, ελεύθερα για να πρέπει να ρυθμιστούν. Ή λέμε ότι δεν αρκεί αυτό που προτείνεται από την Επιτροπή ε, και αυτό ακόμη το οποίο εγώ προσπάθησα να αναδιατυπώσω, μπορεί να πείτε δεν αρκεί. Είναι ελλειπές, λίγο, ανεπαρκές. Έστω. Και τοτε τεστ θα αφήσουμε. Η παράκλησή μόνο προς τους σκιώδεις ηγητές είναι... Εντάξει, για το ECR κατάλαβα και για τους αριστερούς ακόμη, την δηλαδή, κατάλαβα, ούτως ή άλλως μας λέτε όχι. Αλλά θα παρακαλούσα τους και ηγητές να ρωτήσουν στις ομάδες τους να το θέσουν το θέμα. Γιατί με μένα η κυρία Γέρα Σέντερ μου λέει déjà vu, κάποιοι άλλοι μου εκφράζουν και στους ελληνοκράτες ακόμη αφιβολίες για το ότι ε, είναι ε, καλό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν υπάρχει μια πιστική πλειονοψηφία η οποία λέει όχι, θα το σκεφτούμε διαφορετικά. Ιδάλλως να προχωρήσουμε και αυτό θα είναι η αρχή της ιστορίας. Περιμένω λοιπόν τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι θα έρθουν το Δεκέμβριο να τα πούμε, αν έρθουν. Ευχαριστώ. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 30 Δεκεμβρίου, ψηφοφορία στι 11 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή. Ε, γίνεται λόγο για ψηφοφορία στην Ολομέλεια, εντάξει δεν έχουμε φτάσει εδώ ακόμα, αλλά νομίζω θα πάει το Μάρτιο του 2014. Όμως ε, προθεσμία υποβολή τροπολογιών η 30 Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φλακενστάιν. Επόμενο θέμα, τροποποίηση του κανονισμού για τους ε, ταχογράφους για τη συσκευή ελέγχου. Να επενθυμίσω ότι η θέση, η απόφαση του Συμβουλίου ε, δημοσιεύθηκε ε, την 21η Νοεμβρίου και το κείμενο που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επετέφθη μεταξύ εισηγητή και οδών και Συμβουλίου. Ω εκ τούτου, το σχέδιο σύσταση τη κυρία Τσικάου για δεύτερη ανάγνωση δεν συμπεριλαμβάνει τροπολογίε. Ξέρω ότι ίσως να υπάρχουν ζητήματα κατά πόσο κάποιες ομάδες ε, συμφωνούν με τις ε, συμβαστικές ή όχι. Η επιλογή που έχουν είναι να ψηφίσουν υπέρ ή κατά του συμβασμού. Όμως η 12η Νοεμβρίου είναι ε, η προθεσμία. Η κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ψηφισουν υπερ κατα του συμβασμου ομως η 12 η νοεμβριου ειναι η προθεσμια κυρια τσικαου ευχαριστω πολυ προεδρε πρωτα απ ολα θα ηθελα να ευχαριστησω τη Γραμματεία και τους ασκαιώδεις εισηγητές για τις ε, σκληρές προσπάθειες και τη στήριξη που μου παρήχαν καθ' όλη τη διαδικασία τη διαπραγματεύσαμε με το Συμβούλιο. Πάνω από δύο χρόνια ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα. Και πράγματι, το έγγραφο που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή αντικατοπτρίζει τις διαπραγματεύσεις που κάναμε κατά τη διάρκεια τεσσάρων προεδριών του Συμβουλίου. Ως εισηγήτρια θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή Τραν και το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει αυτή τη συμφωνία, καθώς αντανακλά πληρέστατα τις διαπραγματεύσει ε, που κάναμε. Τώρα, επί του περιεχομένου της ε, συμφωνίας, δεν θέλω να επισέλθω στις λεπτομέρειες για τις ε, νέες ε, τεχνικές προδιαγραφές του νέου ψηφιακού τεχογράφου της συσκευή ελέγχου. Προφανώς υπάρχουν νέες βελτιώσεις ε, με επικοινωνία εξ αποστάσεως, ε, δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων και το καθεξής. Ουσιαστικά ζητήσαμε ζητήθηκε μάλλον να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να δεχθούν αυτό το σύστημα της επικοινωνίας εξ αποστάσεως, ώστε να μην είναι μόνο ο κλάδος ε, των μεταφορών που θα πρέπει να επενδύσει στους νέους ε, έξυπνους τεχογράφους νέας γενιάς, αλλά και οι ελεγκτικοί φορείς να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις πληροφορίες ε, που παρέχονται από αυτές τις συσκευέ. Και το Κοινοβούλιο κατάφερε να βελτιώσει τις διατάξεις και την προστασία των δεδομένων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας σε ό,τι αφορά τα δεδομένα τοποθεσίας, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη συμπερίληψη κάποιων και άλλων σημείων πέραν ε, ε, του τόπου ένραξης και λήξης της βάρδιας. Πετύχαμε λοιπόν μετά από τρεις ώρες συνεχούς οδήγησης να ε, καταγράφεται η τοποθεσία. Μετά η χρήση του δορυφορικού σήματος ε, θα γίνεται δωρεάν και οι και ε, συσκευέ ελέγχου θα ε, εισαχθούν εντός 36 μηνών μετά την υιοθέτηση του κανονισμού. Θα κυκλοφορήσουν στην αγορά. αλλά οι 36 μήνες αρχίζουν να τρέχουν μετά από την ε, ε, θέση σε ισχύ. Τώρα, για το ζήτημα ITS, Intelligent Transport System, το κείμενο συμπεριλαμβάνει νέες ε, διατάξεις και είναι σημαντικό το ότι καταφέραμε να εισαγάγουμε διατάξεις σε ό,τι αφορά την τυποποιημένη διαπαθή. Standardized Interface για τα πνευματικά δικαιώματα και την χρήση εξωτερικών συσκευών. Το Κοινοβούλιο επέμεινε και κατάφερε να καταγραφεί στο κείμενο ότι όλα τα φορτηγά από μια ημερομηνία και μετά θα έχουν τέτοιες ευφυείς συσκευές, ούτως ώστε εντός 15 ετών από την εισαγωγή των έξυπνων ταχογράφων όλα τα οχήματα στις διεθνείς μεταφορές να έχουν ε, τέτοια συσκευή. Για τα γραφεία ελέγχου έχει ενισχυθεί ο ρόλος τους ή μάλλον για το προσωπικό ελέγχου. η Επιτροπή έχει νέες προτάσεις για την κατάρτιση των ε, ελεγκτών και συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για την κοινή ερμηνεία της κοινωνική νομοθεσίας. Για τις προσωρινές κάρτες έχουμε ενισχυμένους ελέγχους για τους οδηγούς που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ψηφιακούς ταχογράφους και έτσι ε, ο έλεγχος τους θα γίνεται πιο αποτελεσματικά. Έχουμε βελτιώσει ε, την κατάσταση ότι αφορά τις ευθύνες ε, του κλάδου των μεταφορών. Η πρόταση ε, συγχώνευσης διαφόρων τύπων καρτών και αδειών οδήγησης απερίφθη, γιατί θεωρήθηκε ότι δεν είναι αρκετά όρημη. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική νομοθεσία, το Κοινοβούλιο πραγματικά πάλευσε σκληρά. Και έτσι η νομοθεσία αφορά μόνο τους επαγγελματίες οδηγούς. Ο κανονισμός λοιπόν δεν θα ισχύει για τα φορτηγά κάτω των 7,5 τόνων που μεταφέρουν ε, υλικά εξοπλισμό ή μηχανήματα ε, για τον οδηγό, όμως ε, όταν δεν πρόκειται για επαγγελματία οδηγό. Έχουμε αυξήσει τώρα την ακτίνα από τα 50 στα 100 χιλιόμετρα σε κάποιες περιπτώσεις και θεωρώ συμπερασματικά ότι η πρόταση είναι καλή ακόμα και για τους συναδέλφους στη Γερμανία που προσπάθησαν να υπάρξει αύξηση από τα 100 στα 150 ή στα 200 χιλιόμετρα. Τα 100 χιλιόμετρα που έχουμε τώρα είναι ήδη η διπλάσια απόσταση σε σχέση με το, τα 50 χιλιόμετρα που ήταν στην αρχική πρόταση και έχουμε και την ευρωπαϊκή εξαίρεση που αφορά τους μη επαγγελματίε οδηγούς. Θα μείνω εδώ και καλό τους συναδέλφους να εγκρίνουν τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Να επανθυμίσω στους συναδέλφους ότι στη θέση δεύτερης ανάγνωσης δεν μπορείς να ξαναπαρουσιάσεις τροπολογίες που δεν πέρασαν στην πρώτη ανάγνωση. Δηλαδή, βασικά, το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς με τις τροπολογίες είναι να αποκαταστήσει ε, στο εν μέρη τη θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση. Αν δεν σα αρέσει λοιπόν ε, η θέση που είχε το κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση, δύσκολα τα πράγματα, έτσι είναι τα πράγματα. Ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό και η προθεσμία είναι 28 Νοεμβρίου. Όσοι λοιπόν προσπαθήσουν να καταθέσουν τροπολογίες που δεν αποκαθιστούν τη θέση του Κοινοβουλίου, δεν αποκλειστούν. Θέλει κανείς να πει κάτι, είστε όλοι ικανοποιημένοι με τα σχόλια της με την παρουσίαση της Σιλβίας. Ήθελα απλώ να τον ευχαριστώ για τη δουλειά. Πολύ καλή συνεργασία για τον ηλεκτρονικό ψηφιακό ταχογράφο έστω και αν δεν πέρασαν όλα όσα εγώ θα ήθελα, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ καλά το αποτέλεσμα εν τέλει. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ο κύριος Χέντμπερκ από την Κροπεσιόν. Αν μπορείτε να είστε και σύντομος για να σε ξαναδούμε με καλό μάτι. Μάλιστα, θα είμαι πολύ σύντομα. Φυσικά υποστηρίζουμε το τελικό συμβαστικό κείμενο που συμφωνήθηκε μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στον τριμερή διάλογο και την ακόλουθη πρώτη τη θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου και θα καλωσορίσουμε και μία απόφαση από το Κοινοβούλιο που θα διευκολύνει την ε, ταχεία υιοθέτηση αυτού του σημαντικού κανονισμού. Περί πρόκειται. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το συντομότερο δυνατόν θα έχουμε στην αγορά αυτή τη νέα γενιά τακογράφων γιατί που θα είναι παραβίαστη γιατί αυτό θα έχει και ωφέλη σε σχέση με την οδική ασφάλεια, με την ευημερία των οδηγών και με το να έχουμε ίσους κανόνες ε, για τους ε, επιχειρηματικούς φορείς. Και φυσικά ανυπομονούμε να εγκρίνει το Κοινοβούλιο το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους και εισηγητές ε, για την επικοδομητική τους δουλειά για το φακελό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω για σαφήνεια, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 28 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι και να σας πω ότι η ψηφοφορία θα λάβει η χώρα την Τρίτη στις 17 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την εισηγήτρια, δεν υπάρχει κάτι τίποτα διάφορα. Απλά να σας υπενθυμίσω, εάν χρειάζεται, ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει η χώρα στις Βρυξέλλες 16 Δεκεμβρίου στις 3 το μεσημέρι και θα συνεχίσουμε και στις 17. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Καλό σας βράδυ.